Okay. Good morning to everybody. And I open now our committee meeting for today. Κυρίσω την πανηγυρική έναρξη της συνεδρίασής μας. Πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, μήπως υπάρχει καμία αίτηση, κανένα αίτημα αλλαγής. Όχι. Άρα εγκρίνεται. Δεύτερον, οι ανακοινώσει του Προέδρου. Όπως φαντάζεστε, αναμεταδίδεται η συνεδρίαση. Προσπαθήστε λοιπόν να συμμορφωθείτε με το, με να συμμορφώσετε τη συμπεριφορά σας με τα δέοντα. Έπειτα, έχετε κατάλογο μηνυμάτων, αν θέλετε κανένα αντίγραφο επιστολής, να, ζητήσει, να το ζητήσετε από την γραμματεία. Για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, το τίσα πρώτα, Είχαμε ζητήσει περισσότερη διαφάνεια και στις 10 Μαρτίου το Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει την εντολή διαπραγματεύσεων της ΤΙΣΑ σημαντικό βήμα και αυτό για καλύτερες συνεννοήσεις και συζητήσεις με την κοινωνία των πολιτών και οι πιο λογικές για τις εμπορικές συμφωνίες. Αυτή η δημοσιοποίηση λοιπόν πέντε μήνες μετά ήδη που αποφάσισαν να, και να, δημοσιευτούν και, να δημοσιευτεί και η εντολή για το TTIP είναι από τα πρώτα βήματα για τον αποχαρακτηρισμό τέτοιων εγγράφων και θα έπρεπε να είναι το πρότυπο όλων των εμπορικών διαπραγματεύσεών μας. Να δημοσιεύονται δηλαδή όλες οι εντολές όσο το δυνατόν συντομότερα ώστε όλοι και όλες να γνωρίζουν τι συζητιέται. Έπειτα για την εμπορική συμφωνία Ευρώπης-Σιγκαπούρης. Η παλαιότερη προηγούμενη επιτροπή είχε αποφασίσει την τελευταία μέρα της θητείας της, να προσφύγει στο δικαστήριο για το θέμα της μικτής συμφωνίας για τη Σιγκαπούρη. Η δε νέα επιτροπή το συζήτησε πολύ το πράγμα και στις 4 Μαρτίου επανεξέτασε την απόφαση αυτή και ζήτησε γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως προς το με ποια κριτήρια γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση της Μικτής συμφωνία. Και τέλος, η συμφωνία για το περιβάλλον ΚΟΥΤΣ. Ο πέμπτος γύρος αρχίζει αυτή την εβδομάδα για τα προϊόντα ανάλυσης και παρατήρησης του περιβάλλοντος. Στις 6 Απριλίου η Κομισιόν θα κάνει μια σχετική ανακοίνωση. Εδώ. Ωραία. Αυτά ήταν το σημείο 2. Και τώρα περνάμε στο σημείο 3. Συζήτηση ή ανταλλαγή απόψεων με τον εξοχότατο κατακάμι πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ένωση. Και το θέμα είναι βέβαια οι εμπορικές σχέσεις Ένωσης Ιαπανίας. Πολλές φορές συζητήσαμε την πρόοδο των συνομιλιών και χαίρομαι πραγματικά που είναι εδώ παρόν ο πρέσβης Κατακάμι. Διότι έχω την εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργό Αμπέι έχει φιλόδοξο στόχους, δηλαδή να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις στα τέλη του 2015. Uh, uh, Λίγοι μήνες δηλαδή μόνο απομένουν. Εννέα για την ακρίβεια. Από τον Απρίλιο του 2013 είχαν αρχίσει οι συνομιλίες και, είχαμε πει να παρακολουθούμε τι γίνεται. Προ στιγμή φαίνεται ότι κινούνται καλά οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσει: και μπορεί να έχουν και καλή κατάληξη. Θα δούμε αν τελειώσουν στο τέλος του έτους. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι εμπορικές συμφωνίες για ασφάλεια προέχει της ταχύτητος. Λοιπόν, θα δούμε. Ο πρεσβευτής, στον οποίο δίνω αμέσως το λόγο. Ορίστε κύριε πρεσβευτά μου. and good morning to distinguished members of the European Parliament. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ. Θα κάνω μια εισαγωγική παρουσίαση και μετά είμαι διαθέσιμος για ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, Είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα που έχω την δυνατότητα να μιλήσω στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για τις ε, εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας. Θα ήθελα εδώ να εκφράσω την υψηλή μου εκτίμηση για τον ρόλο τον οποίο παίζεται στην ενίσχυση ε, του διεθνούς εμπορίου της Ένωσης με άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ιαπωνία. Για να δούμε πώς έχουν σήμερα οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ιαπωνία. Και οι δύο εταίροι έχουν ε, εδώ και δεκαετίες συμμερίζονται θα έλεγα κοινέ αξίες όπως το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία. Η σχέση μας έχει αναπτυχθεί με θαυμαστό τρόπο θα έλεγα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει προσφέρει πολλά στον οικονομικό τομέα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Κίνα είναι ο τρίτος εμπορικός εταίρος, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ιαπωνία είναι η έβδομη ε, χώρα ε, όπου καταλήγουν οι ευρωπαϊκές εξαγωγές. Υψηλά ποσά και προς τις δύο κατευθύνσεις σε αιτήσια βάση συνολικά 54 δις ε, ευρώ. Και υπάρχει βέβαια και ένα πλεόνασμα σε επίπεδο εμπορικού ισοζυγίου από πλευράς της Ιαπωνίας οι άμεσες επενδύσεις οι ευρωπαϊκές στην Ιαπωνία είναι θα έλεγα οι περισσότερες από όλους τους εταίρους που επενδύουν στη χώρα μου. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ιαπωνία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη μετά από την Κίνα και την Ηνωμένε Πολιτείες. Υπάρχουν χιλιάδες ε, ιαπωνικές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 500.000 εργαζόμενοι συνολικά. Αυτό έχει οδηγήσει και στην ενίσχυση των πολιτικών και ε, διπλωματικών σχέσεων. Συνεργαζόμαστε σε πολλά θέματα όπως ε, η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή. Υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στις ε, αρμόδιες υπηρεσίες των, της χώρας μου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιοχές όπως το Μαλί. Συνεργαζόμαθα επίσης και στον τομέα της καταπολέμησης της πειρατείας στον Ινδικό ωκεανό. Συμπληρωματικά έχουμε ξεκινήσει και διάλογο και στον τομέα της, ε, ε, των κυβερνοεπιθέσεων και στον τομέα των διαστημικών. Έχουμε ενισχύσει γενικότερα και τη συνεργασία μας σε τομείς όπως η πρόληψη των καταστροφών και η καταπολέμηση του ιού έμπολα. Βλέποντας λοιπόν την ολοένα διαβινόμενη σχέση ανάμεσά μας, ένα από τα θέματα τα οποία έρχονται στην επικαιρότητα είναι ο καθορισμός ενός πλαισίου για στενότερη οικονομική συνεργασία μέσα του EPA του FDA. Η προώθηση των εταιρικών σχέσεων με άλλες χώρες είναι σημαντικό θα έλεγα, σημαντικό στόχος της ε, νέας οικονομικής πολιτικής της χώρας, των λεγόμενων Abenomics με το όνομα, από το όνομα του Πρωθυπουργού. Γενικά, ε, οι, εξελίσσονται οι υποθέσεις που μας ενδιαφέρουν, αλλά όχι ίσως με την ταχύτητα που θα επιθυμούσαμε. Το FDA, ας πούμε, δεν είναι μόνο σημαντικό για να αυξηθεί το εμπόριο ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και για συνεργασία σε άλλους τομείς. Βλέπουμε ότι το κέντρο της ε, οικονομικής ισχύω του πλανήτη φεύγει από τη Δύση και πηγαίνει περισσότερο προς την Ασία και γι' αυτό ε, υπάρχει ανάγκη να συνεργαστούμε ακόμα στενότερα στον τομέα της οικονομίας, στον τομέα της, ε, των κανόνων της αγοράς. Η ολοκλήρωση του EPA-FDA με την Ιαπωνία θα είναι κινητήρια δύναμη και για τις δύο πλευρές. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι έχει σημασία να υπάρξουν απτά ωφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας το ταχύτερο δυνατόν και στο ευρύτερο δυνατό επίπεδο. Είναι ενθαρρυντικό λοιπόν ε, που η συνάντηση Άμπε και Γιούγκερ ε, έδειξε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμφωνία ε, καταρχάς σε σχέση με το EPA-FDA. Ε, θα υπάρξει σημαντική πρόοδος λοιπόν το 2015. Η Επίτροπος Μάλστρομ είχε επιτυχείς συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας και τον Υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας. Πιστεύουν ότι το χρονοδιάγραμμα είναι φιλόδοξο μεν, αλλά εφικτό και θα πρέπει να συνεχιστούν και να εντατικοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι ήταν λοιπόν μια καλή αρχή για να μπορέσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία επί της αρχής. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν για η ε, FDA έγιναν στις Βρυξέλλες ε, τον προηγούμενο μήνα. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία, 180 ε, μελών με πολλούς εμπειρογνώμονες από πάρα πολλούς τομείς του δημόσιου τομέα στην Ιαπωνία. Έμαθα ότι σε ορισμένους τομείς οι διαφορές έχουν ξεκαθαριστεί περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν. Είναι πολύ φυσικό θα έλεγα να υπάρχουν διαφορές στα πλαίσια μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας. Νομίζω ότι είναι μια θετική πλευρά αυτή, γιατί δείχνει ότι έχουμε περάσει στις πραγματικές διαπραγματεύσεις, όπου θα υπάρξουν πολύ παραγωγικές συζητήσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια του ενάτου γύρου των διαπραγματεύσεων συζητήσαμε πάρα πολλούς τομείς όπως πρόσβαση στην αγορά αγαθών, υπηρεσιών, επενδύσεις, MTMs και ε, προμήθειες. Στα πλαίσια αυτού του γύρου οι διαπραγματευτές και των δύο πλευρών νομίζω ότι πέτυχαν καλά αποτελέσματα εντοπίζοντας ε, τις δυσκολίες και πιστεύοντας ότι θα υπάρξει αυτή η συμφωνία υψηλού επίπεδου. Συνειδητοποιώντας βέβαια και τις διαφορές. Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία επί της αρχής μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πρέπει όπως είπαμε να συναντώμεθα σε ε, δίμηνη βάση και να συνεχίσουμε και τις επιπλέον επαφές όπου αυτές είναι απαραίτητες. Νομίζω ότι είμαι σε θέση να δώσω κάποιες λεπτομέρειες τώρα για τις διαπραγματεύσεις. Για τα μη δασμολογικά μέτρα. Έχουμε σαφώς προχωρήσει στην εφαρμογή των ε, δράσεων ε, στις οποίες είχαμε καταλήξει μετά την έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων. Έχουμε προωθήσει και άλλα θέματα αν και βέβαια δεν θα εφαρμοστούν όλα αυτά πλήρως αν δεν κλείσουν οι διαπραγματεύσεις. Τα δύο τρίτα των θεμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στον ενδιάμεσο οδικό χάρτη έχουν ήδη αντιμετωπιστεί και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμεθα και στα υπόλοιπα θέματα. Για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας η Ιαπωνική κυβέρνηση μέχρι τώρα συνεχίζει να υιοθετεί ε, τον κανονισμό της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών. Συνεργάζεται επίσης ε, η Ιαπωνία με τις υπόλοιπες χώρες για το IWVTA, για το σύστημα έγκρισης τύπου, παγκόσμιο σύστημα έγκρισης τύπου αυτοκινούμενων οχημάτων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα διευκολύνει κατά πολύ τις δραστηριότητες, θα υπάρξει ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης για το σύνολο του οχήματος. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω λίγο και για τους σιδηροδρόμους. Υπάρχουν ε, τρεις ιδιωτικές ε, ε, ιαπωνικές επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, σιδηροδρόμων, ε, οι οποίες προμηθεύονται από όλο τον κόσμο εξοπλισμό. Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες στην αρχή των διαπραγματεύσεων, αλλά έχει επιβεβαιωθεί ότι οι προμήθειες θα πρέπει να γίνονται από εδώ και πέρα με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της έλλειψης διακρίσεων και οι εταιρείε αυτές, οι επιχειρήσεις αυτές, οι σιδηροδρομικές έχουν δώσει πολλές, έχουν δημοσιοποιήσει ε, τις προμήθειές τους. Ε, υπάρχουν επιχειρήσεις που θέλουν να ε, χρησιμοποιήσουν την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και τον ε, τεχνολογικό ευρωπαϊκό εξοπλισμό. Υπήρξαν επαφές σε επίπεδο επιχειρηματικό και στο Μιλάνο και στη Λίλ και στην Γερμανία, στο Ντίσσελντορφ. Εκεί εξηγήσαμε ποιες είναι οι μελλοντικές μας δράσεις και προβλέψεις στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων λοιπόν θα εντατικοποιηθεί ο διάλογος ανάμεσα στη σιδηροδρομική βιομηχανία της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ήδη υπάρξει επαφές όπως είπα ε, στις επαφές αυτές έχουν πάρει μέρος πάνω των 100 εμπλεκομένων ε, και από την πλευρά των κατασκευαστών και από την πλευρά των χρηστών, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων δηλαδή. Εμείς προσπαθούμε να εμβαθύνουμε την αμοιβαία κατανόηση, την συνεργασία και τις ανταλλαγές ανάμεσα στους εταίρους. Ε, νομίζω ότι αυτό θεωρήθηκε ιδιαίτερα θετικό από τους συμμετέχοντες και των δύο πλευρών. Η Ιαπωνική κυβέρνηση λοιπόν θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον σιδηροδρομικό λεγόμενο διάλογο. Πέρα λοιπόν από τις προμήθειες των τομέα των σιδηροδρομικό ε, ασχολούμεθα και με τις ανησυχίες που εκφράσατε ε, για αυτούς τους τομείς στο παρελθόν. Ε, σε άλλους τομείς τα πράγματα παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο και δεν μπορεί να υπάρξει κάποια βελτίωση εάν δεν ολοκληρωθεί και εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία. Συνεπώς λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία πρέπει να αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες τις διαφορές τους. Είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Νομίζω ότι το EPA-FDA θα δημιουργήσει ε, πάρα πολλά ωφέλη για τον μέγιστο δυνατό αριθμό πολιτών. θα πρέπει να δούμε τα μόνιμα ωφέλη τα οποία θα δημιουργήσει η συμφωνία αυτή ευρύτερα. Η φωνή της Ευρώπης και της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών και των κυβερνήσεων ακούγονται βέβαια και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι θα ευγνώμονες λοιπόν για, για τη συνέχεια των προσπαθειών τις οποίες κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πεπισμένος ότι η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρουν τα απαιτούμενα μέτρα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Ελπίζω να συνεχίσουμε την συνεργασία μας για να πετύχουμε τον στόχο μας. Thanks a lot, uh, ευχαριστούμε πρεσβευτά και όντως κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε προκειμένου να πετύχουμε μια καλή συμφωνία. Τώρα, να δώσω το λόγο στο μόνιμο εισηγητή μας και μετά στους σκιώδες εισηγητές. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τον ε, πρεσβευτή Κατακάμι, τον οποίο πάντα δεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά εδώ. Σας ευχαριστώ για τις απόψεις που μας παρουσιάσατε για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Έχουν περάσει δύο χρόνια από την έναρξη των ε, διαπραγματεύσεων. Η αναθεώρηση του πρώτου έτους ήταν θετική, αλλά τώρα συνεχίζονται οι συζητήσεις και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Προσδευτά, έχει παρουσιάσει ένα νέο κατάλογο μη δοσμολογικών φραγμών που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει από πλευρά της Ιαπωνίας και αυτό ήταν σαφές και στην αναθεώρηση τη μονοετή. Ωστόσο θα ήθελα να σχολιάσετε τον δεύτερο αυτό κατάλογο μη δασμολογικών φραγμών και τον τρόπο που η Ιαπωνία αντιμετωπίζει την ανάγκη επίλυσης των ζητημάτων αυτών. Για να σας το πω ανοιχτά, αυτό που θέλω να μου πείτε είναι ποια είναι η άποψη πραγματικά της Ιαπωνίας για την ρεαλιστική προσέγγιση των διαπραγματεύσεων. Τι σημαίνει ακριβώ αυτό. Καταλαβαίνω τα σχόλια που κάνατε και είπατε ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις των συντομότερων δυνατών. Φέτος, κατά πάσα πιθανότητα. Όλοι αυτό το στόχο έχουμε. Αλλά, τι σημαίνει η ρεαλιστική αυτή προσέγγιση. Η Ιαπωνία εξετάζει το δεχόμενο να υπάρξει μια γενική μόνο συμφωνία λιγότερο φιλόδοξη και να αναβληθεί για μετέπειτα φάση η ρύθμιση άλλων λεπτομερών ζητημάτων όπως τα κανονιστικά ζητήματα. Μήπως διακυβεύουμε έτσι να υπονομεύσουμε μία σημαντική και πραγματικά ωφέλιμη συμφωνία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τις οικονομίες αμφότερων των πλευρών να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, αλλά θέλουμε να είναι και καλή και ισορροπημένη αυτή η συμφωνία. Και φυσικά αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της ιαπωνικής πλευράς σε ό,τι αφορά τις δεσμολογικές ε, πτυχές των φραγμών αλλά τα ζητήματα αυτά, τα αριθμιστικά ζητήματα, ακόμα και ενός ε, είδους διακριτικής μεταχείρισης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να επιληθούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Θα γίνει λοιπόν μια πολύ σημαντική σύνοδος το Μάιο. Έχουμε ακόμα δύο ευκαιρίες σε έναν ε, ενδιάμεσο γύρο διαπραγματεύσεων και σε έναν επίσημο γύρο διαπραγματεύσεων όπου και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε θετικές εξελίξεις ε, πριν τη Σύνοδο, προκειμένου να υπάρχει μια σαφή εικόνα και να καταδείξουμε ότι συνεχίζουμε να ε, επιδιώκουμε τον στόχο μιας φιλόδοξης και σημαντικής συμφωνίας και για τις δύο οικονομίες. Κατά δεύτερον, ε, πρεσβευτά. Να σας ρωτήσω, Μπορούμε να υπολογίζουμε στη δέσμευση της Ιαπωνίας στις διαπραγματεύσεις αυτές. Γνωρίζοντας ότι η Ιαπωνία διεξαγάγει και άλλες πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του TPP. Κάποιοι στην Ευρώπη ενδεχομένω να θεωρούν ότι είναι τόσο περίπλοκο το θέμα του TPP που ενδεχομένω να είναι σε πιο υψηλή θέση στις προτεραιότητες και στην ατζέντα της ιαπανικής πλευράς. Θα θέλαμε λοιπόν να μας επιβεβαιώσετε ότι η Ιαπωνία κάνει τα δέοντα για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα των διαπραγματεύσεων με την Ευρώπη. Προκειμένου να υπάρχει, όπως σας είπα, μια φιλόδοξη και πραγματικά ωφέλιμη συμφωνία με την Ευρώπη. Θα ήθελα επευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι κάναμε, διοργανώσαμε για την επόμενη Τρίτη μία συνάντηση για, με την αντιπροσωπεία για τις, για τις σχέσεις με την Ιαπωνία, να συζητήσουμε θέματα όπως η σειροδρομή μεταξύ άλλων. Θέλουμε να ακούσουμε τις ανησυχίες και της Ιαπωνικής πλευράς και της Ιαπωνικής βιομηχανίας. Έχουμε ήδη ακούσει τις ε, παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά τις πραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήλθατε εδώ, κύριε Πρεσβευτά, για τα σχόλιά σας, τις εξηγήσεις σας και αυτές τις δύο ερωτήσεις ήθελα να σας θέσω, να ακούσω και ποια είναι η απάντησή σας, για να γνωρίζουμε πόσο μπορούμε να πιστεύουμε στην σύναψη μιας καλής συμφωνίας φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα ο κύριος Βαλέσα από το είναι ο Ινέος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρεσβευτά, όπως ξέρετε, η προστασία των καταναλωτών είναι ύψης της σημασίας θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 89 έχουμε θέσει την απέτηση όλα τα τρόφιμα να φέρουν επισήμανση για την ε, παρτίδα παραγωγής και έχουμε προβλέψει και σχετικές κυρώσεις αν αυτό δεν γίνεται σεβαστό. Στην Ιαπωνία αυτή η κωδική λάτ δεν είναι υποχρεωτική, παρόλα αυτά τα συστήνει αυτά, τη συστήνει τη χρήση του στο Υπουργείο Υγείας ε, και Γεωργίας. Αυτό σημειώθηκε και το 2014 και έχει τεθεί ως θέμα και σε οκτώ εμπορικές συμφωνίες μεταξύ άλλων και από την Ένωση Εξαγωγών Ινοπνευματοδών της Ιαπωνίας. Χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός ε, από πλευράς της Ευρώπης ε, όταν πρόκειται για εξαγωγές προς την Ιαπωνία και αυτό ε, διευκολύνει την ανείχνευση, τον εντοπισμό των προϊόντων για να περιορίζεται ο κίνδυνος στην υγεία των καταναλωτών. Δυστυχώς ε, υπάρχουν κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα με διαγραμμένο τον κωδικό αυτό. Και αυτό φυσικά πλήττει και την ε, εμπιστοσύνη των προϊόν και την εμπιστοσύνη των ε, πολιτών στην επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που χρειάζεται. Η κυβέρνηση λοιπόν της Ιαπωνίας σκέφτεται να εφαρμόσει νομοθεσία, να περάσει νομοθεσία προκειμένου να προαπαιτείται η επισήμανση των προϊόντων με τον αρχικό κωδικό ΛΑΤ σχετικά με την παραγωγή τους. Και να δράσει σε περίπτωση που υπάρξει παραποίηση των κωδικών αυτών. Έχει διαγραφεί ο κωδικός αυτός. Μας δώσατε, ξέρετε, τον κατάλογο των προτάσεών σας και αυτό που πραγματικά ρωτάω είναι κατά πόσο θα ήσασταν διτεθειμένοι να επεκτείνετε τον κατάλογο αυτό και σε περίπτωση που είσαστε διτεθειμένοι τι θα συμπεριλαμβάνονταν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καμάλα από το ECR δεν είναι εδώ, ο κύριος Λάμπσδορφ ούτε αυτός παρίσταται. Ο κύριος Σόλτς λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρα και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον κύριο Πρεσβευτή για τις εξηγήσει σε ό,τι αφορά το πώς έχουν τα πράγματα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρώπης για την εμπορική συμφωνία. Θα ήθελα από πλευρά της ομάδας μου να υπογραμμίσω με σαφήνεια ότι είμαστε σαφώς υπέρ μια εταιρική σχέση για τις κοινωνικές διαπραγματεύσεις με ίδια πρότυπα και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα συμφέροντα της Ιαπωνίας αλλά και των 28 κρατών μελών των λαών αυτών λοιπόν. Θα πρέπει να με τη βάση των συμφερόντων αυτών να αξιολογήσουμε και την, την τρέχουσα κατάσταση και συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο ότι η ποιότητα προηγείται της ταχύτητας. Θα πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε δηλαδή ποιος είναι ο απότερος στόχος της συμφωνίας, τι θέλουμε να πετύχουμε πώς θέλουμε να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας. Τέσσερις, τέσσερις ερωτήσεις και προς τον πρεσβευτή και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως που θα πάρει μέρος φαντάζομαι στη συζήτησή μας. Κατά πρώτον, πώς έχει σήμερα η κατάσταση των διαπραγματεύσεων σε σχέση με τον, τη συμφωνία μεταξύ των ΙΠΑ και των κρατών ε, από την άλλη πλευρά του ειρηνικού μεταξύ άλλων και της Ιαπωνίας. Νομίζω ότι αυτό το θεωρεί προτεραιότητα η Ιαπωνία το 2015 και τίφονται και θέματα οικονομικής συνεργασίας ε, των ε, χωρών του ειρηνικού. Αυτό φυσικά επηρεάζει και τις διμερεί διμερείς ε, διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας αλλά και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΙΠΑ πλαίσια του TTIP, το είπε και ο εισηγητής αυτό. Αυτές οι διαπλοκές λοιπόν θα ήθελα να διαφωτιστούν από πλευράς της Ιαπωνίας. Δεύτερη ερώτηση και συνδέεται με την πρώτη ερώτηση. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει πραγματική δυνατότητα να υπάρξει κανονιστική συνεργασία με μορφές που θα έχουν συμφωνηθεί που θα λάβουν υπόψη τις ε, πολύ διαφορετικές παραδόσεις σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο και σε ό,τι αφορά το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά την Ιαπωνία. Αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν. Είπατε κύριε Πρεσβευτά ότι κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων είναι σαφές το που Έγινε οι διαφορές. Δώστε μας λοιπόν ένα-δύο παραδείγματα. Πού βρίσκονται ακριβώς οι διαφορές. Τρίτη ερώτηση. Μία ερώτηση να σας κάνω για το κατά πόσο η Ιαπωνία έχει μια άποψη για τη συμπερίληψη του ESDS στην ε, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Να μας πει τη γνώμη της σε ό,τι αφορά δηλαδή, την επίλυση διαφορών δημοσίου και δυτικού τομέα. Τελευταία ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε κάτι από ιαπωνικής ε, άποψης για το κεφάλαιο βιωσιμότητας εμείς θέλουμε να υπάρχουν σαφής και δεσμευτική συμπερίληψη όλων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ε, πτυχών. Ποια είναι η στάση της Ιαπωνίας και αυτό το ερωτώ και ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θα ήθελε να τοποθετηθεί. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, ο κ. Μπουκνέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς, ε, κύριε Πρεσβευτά για την συνομιλία αυτή, για την ευκαιρία που μας δίνεται να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με τις ερωτήσεις του κυρίου Σόλτς. Να θέσω το θέμα του ESDS. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό το θέμα για σας κύριε Πρεσβευτά. Πολύ σημαντικό και πώς έχουν ε, οι διαπραγματεύσεις στο σημείο αυτό. Κατά δεύτερον, είμαστε πολύ επικριτικοί σε ό,τι αφορά τις αρνητικές λίστες, τις αρνητικές, τους αρνητικούς καταλόγους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, γιατί είναι δύσκολο να γίνουν μετέπειτα διαπραγματεύσεις και προσαρμογές όταν υπάρχουν ε, αρνητικοί κατάλογοι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ε, υπηρεσίες. Ποια είναι η άποψή σας. Τρίτη ερώτηση. Είπατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, ότι κάποια πρόσθετα στα τρόφιμα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, τα οποία έως τώρα ήταν απαγορευμένα στην Ιαπωνία λόγω των κινδύνων που επιφέρουν στην υγεία. Στην Ιαπωνία είχατε πολύ υψηλά πρότυπα στον τομέα αυτό. Τι σας επηρέασε λοιπόν για να αλλάξετε την τοποθέτησή σας αυτή. μήπως ε, με τις διεθνείς συνθήκες και ιδιαίτερως με το TPP προκύπτει μία εξομοίωση με τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή και μία μείωση των προτύπων σε ό,τι αφορά τη χρήση προσθέτων στα τρόφιμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Δύο ακόμα άτομα ζητούν το λόγο. Ο κύριος Φίσας και η κυρία Ρεντίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον πρέσβη κύριο Κατακάμε για την παρουσίασή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη και φιλόδοξη συμφωνία με συγκεκριμένα μέτρα, με κατάργηση των μέτρων που δημιουργούν διακρίσεις που θα επιτρέψει το άνοιγμα της Ιαπωνικής αγοράς κάποια επιμέρους σημεία. Το θέμα των γεωργικών προϊόντων. Νομίζω ότι η προσφορά της ιαπωνικής πλευράς δείχνει μια κάποια έλλειψη φιλοδοξίας ε, και δεν αναφέρομαι σε θέματα όπως ε, τα γαλακτοκομικά, το βόλιο κρέας, το χείριο κρέας, αλλά και στα υποπροϊόντα τους. Στόχος μας είναι να επιτρέψουμε, ορισμένα, να επιτρέψουμε την εφαρμογή ορισμένων μέτρων όπως στα πλαίσια της συμφωνίας με την Αυστραλία ή όπως η συμφωνία της Ιαπωνίας με τις Ηνωμένε Πολιτείες σε τομείς όπως τα αμπελοϊνικά. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις που πρέπει να υπάρξουν και στο, να γίνουν και στον τομέα της, ε, ε, του, χαρακτηρισμού των προϊόντων ονομασίας προέλευσης. Μέχρι τώρα έχουν γίνει μόνο κάποια πρώτα μικρά βήματα, πρέπει να ολοκληρωθούν και να μεγεθυνθούν. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί και μια ρήτρα η οποία στη συμφωνία η οποία θα ε, διασφαλίζει ε, την συμβατότητα των περιοχών ε, ονομασίας προέλευσης με τα διπλώματα ευαισθητεχνίας όπως επίσης και τα δικαιώματα που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ποιες είναι οι σχέσεις, η διασύνδεση μεταξύ των δικών μας συνομιλιών και άλλων όπως και Υπάρχουν συνδυασμοί, συνέργειες. Προσπαθούμε πράγματι να δημιουργήσουμε διεθνή πρότυπα ή έχετε την εντύπωση ότι αυτές οι διάφορες διαπραγματεύσεις καμιά φορά είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Θα με διέφερε ιδιαίτερα να ακούσω τι φρονείτε για την πρόοδο των συνεννοήσεων για τις τηλεπικοινωνίες και τα αυτοκίνητα. και για το ΙΤΑ εμπόριο όπου η Ιαπωνία είναι λιγότερο ανταγωνιστική από την Ευρώπη. Τώρα η Κομισιόν, ο επικεφαλής μάλιστα των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ για την δυνατότητα να σας ενημερώσω. Θα είμαι σύντομος γιατί περιμένετε τις απαντήσεις του Ιάπωνα πρέσβη. Μας υπενθύμησε τις, ε, τα αποτελέσματα της προσπάθειας ε, την οποία κάναμε τον τελευταίο χρόνο. Νομίζω ότι μια πρώτη συμφωνία ήταν μια καλή συμφωνία. Έχουμε ένα πακέτο που παρουσιάζει πλέον εκτήματα και για τον τομέα της αγοράς και προμήθειας ιδιοδρομικών εξοπλισμών. Κάναμε σημαντικά βήματα προόδου και στον τομέα της ανταλλαγής αγαθών. Mr. Chairman, you have recalled the um, Ιδιαίτερα στον τομέα της κατάθεσης πρώτων προσφορών νομίζω ότι ε, έχουμε κάνει θετικά βήματα. Όπως είπε ε, και ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας πρέπει να κλείσουμε στο τέλος του χρόνου. Τι θα γίνει μέχρι τότε. Καταρχάς περισσότερα για τα μη δασμολογικά μέτρα όπως μας υπενθύμησε ο μιλητής, ο εισηγητής ε, και για τον τομέα των δημοσίων προμηθειών πέρα από την διαφάνεια πρέπει να διασφαλίσουμε την δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές ε, και στον δασμολογικό τομέα κάποια πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι στα πλαίσια της πρώτης προσφοράς ε, ε, φτάνουμε στο 85% του ύψους των δασμών, αλλά δεν είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Καλό είναι, αλλά δεν είναι αυτό που επιθυμούμε. Στον τομέα των υπηρεσιών είμαστε αρκετά δεκτικοί και εμείς και οι Άπωνες, αλλά πρέπει κάποια να διευκρινιστούν όπως η ιδιαίτερη, η ιδιόμορφη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα Ιαπωνικά ταχυδρομεία. Η Ιαπωνία δεν έχει εμπόδια στις επενδύσεις, αλλά επίσημα τουλάχιστον, αλλά έχει χαμηλό επίπεδο ξένων επενδύσεων και αυτό ανησυχεί την Ιαπωνική κυβέρνηση. Θα ήθελε η ξένη οικονομία, η μη Ιαπωνική ρευστότητα να έρθει και στη χώρα του. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο σημαντική τομεί με τους οποίους ασχολούμεθα. Φυσικά πολλά υπάρχουν που μένει να γίνουν ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες, ίσως σε κάποιες από τις μεγαλύτερες ε, ε, παγκόσμιες οικονομίες. Αναφερθήκατε στη Συμφωνία Ιαπωνίας-Αυστραλίας. Ε, ε κοιτάξτε, οι διαπραγματεύσεις οι δικές μας προχωρούν αλλά μπορεί να έχουμε μια διαφοροποίηση στα πρότυπα που επιδιώκουμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μια καλύτερη συμφωνία από αυτή που υπογράψαμε με την Κορέα και με την Κίνα, που είναι και οι δύο συμφωνίες βέβαια φιλόδοξες, συμφωνίες του 21ου αιώνα. Αν το Ιαπωνικό πρότυπο είναι η συμφωνία τους με την Αυστραλία και την Ελβετία, αν λέω, ε, γιατί οι συμφωνίες αυτές είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξες από τη συμφωνία ας πούμε με, την, με τον Καναδά. Τέθηκε και το θέμα του TIP. Νομίζω ότι όταν ολοκληρωθεί θα βοηθήσει εφόσον καταφέρει να ανυψώσει το επίπεδο της φιλελευθεροποίησης του εμπορίου στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Αυτό θα είναι κάτι το πάρα πολύ καλό και για την ευρωπαϊκή πλευρά. Το θέμα είναι δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του TIP. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα απασχολήσει και τους Ιάπωνες και νομίζω ότι και ε, η Ιαπωνική ε, διοίκηση, η Ιαπωνική κυβέρνηση θα μπορέσει να ασχοληθεί με όλα αυτά σε ε, μικρό χρονικό διάστημα. Ο χρονισμός μας από εδώ και πέρα πρέπει να ολοκληρωθεί το 15 όπως είπε και ο πρέσβης Κατακάμι. Ε, εγώ πιστεύω σαν κύριος διαπραγματευτής ότι μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά για να το πετύχουμε πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Εμείς αυτή τη γραμμή ε, ακολουθούμε. Αν μπορούμε να το πετύχουμε θα το επιδιώξουμε. Αλλά όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η ουσία και όχι η ταχύτητα. Καλώς, ο κύριος Κατακάμι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Uh, uh, Ήδη από τον uh, Δεκέμβριο, πριν από τον 8ο γύρο των διαπραγματεύσεων, ξεκίνησαν οι συζητήσεις, κατατέθηκε ένας κατάλογος με τα θέματα που περιλαμβάνουν και τεχνικές λεπτομέρειες και προκάλεσε ο κατάλογος αυτός εντατικές διαπραγματεύσεις και στα πλαίσια μάλιστα ε, ε, ενός ιδιαίτερως επικοδομητικού κλίματος. Ε, εγώ λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε στα πλαίσια αυτά και για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, για την ε, πραγματιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων σε αντιπαράθεση με μια πιο φιλόδοξη ίσως ε, αντίληψη. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ιαπωνία σαν παράδειγμα έχει ένα σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Προσπαθούμε εμείς να καταστήσουμε το σύστημά μας αυτό σύμβατο έτσι ώστε να καλύψουμε και τις απόψεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να σταθούμε με πραγματιστικό τρόπο απέναντι στις διαφορές και προσπαθούμε ταυτόχρονα όμως να επιδιώκουμε πολύ φιλόδοξους στόχους που να καλύπτουν μια τέτοια συμφωνία εμπορική για τον 21ο αιώνα. Τώρα, ε, λέγοντας ότι θα τελειώσουμε το 2015, πολλοί μας κατηγορούν ότι βιαζόμαστε να το κλείσουμε για να μειώσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας της συμφωνίας αυτής. Αυτό το διαψεύδω. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ιδιαιτέρως φιλόδοξοι. Συνεχίζοντας όμως χωρίς καθυστέρηση τις διαπραγματεύσεις για το TTIP. Έχουν υπάρξει αρκετές συζητήσεις. Ήδη εξ αρχής όταν ήρθα στις Βρυξέλλες άκουσα πολλές απόψεις που έλεγαν ότι η Ιαπωνία ίσως να δίνει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι ε, έπρεπε στο TTIP. Ε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς δίνουμε εξίσου σημασία και στην, ε, στη συμφωνία αυτή και στη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας. Προφανώς υπάρχει αλληλοεπίδραση. Ξέρετε ότι στα πλαίσια του TTIP έχουν τερματιστεί σε, σε αυτή τη φάση οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχει μια κάποια συνέργεια ανάμεσα στις χώρες μας και υπάρχουν διαφορετικές πλευρές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έχω την ε, αίσθηση όμως ότι αν το TPP συνεχιστεί ε, οι διαπραγματεύσεις, αυτό θα επηρεάσει πολύ θετικά τις δικές μας διαπραγματεύσεις. Να έλθω τώρα στις τελευταίες ε, παρατηρήσεις που έγιναν και από τον εκπρόσωπο των διαπραγματευτών. Για το TPP απάντησα, τέθηκε ένα θέμα για την συνεργασία σε επίπεδο νομικό διακανονιστικό. Προφανώς πρέπει να υπάρξει σωστή συνεργασία στα πλαίσια της συμφωνίας που θέλουμε να υπογράψουμε. Μιλάμε για μια κάποια μορφή εναρμόνισης των νομικών σχημάτων και πλαισίων. Ε, θα πρέπει να πούμε όμως ότι πάνω από τις διαπραγματεύσεις αυτές είχαμε με την ε, δημοσιεύσαμε ένα, ε, μια κοινή ανακοίνωση ε, ανάμεσα στα αρμόδια Υπουργεία της Ιαπωνίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μια πρόταση συμφωνίας για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, για θέματα θεσμικά. Είναι καλό να συνεργαζόμαστε γιατί έχουμε να κάνουμε με δύο ιδιαίτερα προχωρημένες κοινωνίες που ενδιαφέρονται και για το περιβάλλον και για τις νομικές ρυθμίσεις. Το ISDS είναι ένα θέμα το οποίο ε, παρουσιάζει ενδιαφέρον και για σας. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο σύστημα είναι η τελευταία καταφυγή των ε, ε, επενδυτών και μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των επενδύσεων. Εμείς σε όλες τις ε, επενδυτικές συμφωνίες προβλέπουμε κάτι το αντίστοιχο. Ταυτόχρονα έχει σημασία και το συνειδητοποιούμε αυτό να μην υπάρχουν καταχρήσεις από πλευράς των επενδυτών τέτοιου είδους σχημάτων ε, και αυτό να λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων των κρατών μελών. Πρέπει να υπάρξει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των κρατών από τη μία και των επενδυτών από την άλλη. Η συζήτηση που γίνεται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εδώ στην Επιτροπή σας, στα πλαίσια αυτού του συστήματος δηλαδή διαιτησία σε περίπτωση επενδυτικών διαφορών. Είναι κάτι το οποίο θα λάβουμε υπόψη μας και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων ε, για την εμπορική μας συμφωνία. Τώρα για τη βιωσιμότητα, τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντολογικά τα συζητούμε και αυτά και υπάρχει διάλογος με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Ταυτόχρονα πρέπει να είμαι ειλικρινής. Αυτά είναι καινούργια για μας. Η Ιαπωνία δεν διστάζει καθόλου να τα συζητήσει, αλλά και μάλλον Έχουμε δημόσια συζήτηση και διάλογο με τους εκπροσώπους των κοινωνιών των πολιτών όπως σας είπα και με διεθνείς οργανώσεις για αυτά. Ο αρνητικός κατάλογος τώρα, για τον αρνητικό κατάλογο, το μόνο που μπορώ να πω γενικά είναι ότι τον εφαρμόζουμε δηλαδή σε σύγκριση με τον θετικό είναι πιο πολύ, τάσεται πιο πολύ υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Τώρα τα πρόσθετες στοιχεία ε, ε, ουσίες στα τρόφιμα. Φυσικά η ασφάλεια των τροφίμων είναι από τα πιο λεπτά και ενδιαφέροντα θέματα στην Ιαπωνία και φυσικά βέβαια δεν θα επιτρέψουμε τέτοια αλόγιστη χρήση πρόσθετων. Uh, I Εξάλλου, ο κατάλογος των διεθνών ουσιών που χρησιμοποιούνται για, ως επιπρόσθετα στα τρόφιμα από 44 τέτοιες ουσίες, ήδη τις 40 τις έχουμε ταυτίσει και εμείς και απαγορεύσει. Για τους δασμούς για τα γεωργικά, έχει ακουστεί ότι η Ιαπωνία δεν έχει κάνει τίποτα σημαντικό, αλλά εμείς βασικά ως θέση έχουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη της ευαισθησίας, τον ευαίσθητο χαρακτήρα ορισμένων προϊόντων, δεν έχουμε παραλείψει καμία διαπραγμάτευση. Αλλά επειδή βρισκόμαστε στη μέση ορισμένων τέτοιων δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Αν θέλετε θα σας αναφέρω στο μέλλον τα συμπεράσματα. we basically system, Σύμφωνα με το σύστημα των Abenomics που σας έλεγα πριν, έχουμε ταυτίσει, έχουμε βάλει την ένδειξη γεωγραφικής προέλευσης ήδη γιατί προσπαθούμε να βρούμε δημιουργικούς αλλά και ρεαλιστικούς τρόπους για να ικανοποιήσουμε όλες τις πλευρές. Για το TTIP νομίζω τα είπα. Για την αυτοκινητοβιομηχανία, το ΙΤΑ, εμπόριο και τις τηλεπικοινωνίες. Για τα αυτοκίνητα τα ξέρετε όλα. Από 46 πρότυπα τα 37 ήδη έχουν λυθεί και θα συνεχίσουμε να το προσέχουμε. Δεν βλέπω κανένα μεγάλο πρόβλημα ούτε για τις τηλεπικοινωνίες ούτε για το ΙΤΑ εμπόριο. Υπάρχουν τα ίδια υψηλά πρότυπα και στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία. για το αριθμητικό σύστημα ταύτισης. Το παρακολουθούμε και αυτό και η χνηλασιμό θα την εξηγήσω με γραπτός καλύτερα. Αλλά έχουμε σύστημα χνηλασιμότητα μέχρι την πηγή. Αλλά για το BIN, το Batch Identification Number, Προσπαθούμε και αυτό να το εφαρμόσουμε σύμφωνα σε συνεννοήσεις με τους Ευρωπαίους παραγωγούς για να ξέρουμε πού ακριβώς πρέπει να γίνεται η ταύτιση στην Ιαπωνία ή στο εξωτερικό. Ελπίζω να απάντησα, ίσως όχι όλες τις ερωτήσεις, αλλά τις περισσότερες και σας κατευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρεσβευτά. Να ζητήσω από τον εισηγητή αν θέλει το λόγο για να κλείσει η συζήτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέσβη για τις εξηγήσει τις οποίες μας έδωσε. Αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι μια συμφωνία ουσίας και φιλοδοξίας. Μπορούμε να το πετύχουμε και φυσικά περιμένουμε να ξεκινήσει με πολύ ενδιαφέρον ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων, ο οποίος να είναι καθοριστικός. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την συμμετοχή. Uh, Σας ευχαριστώ και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη, το σημείο 3. Επόμενο θέμα, το υπαριθμό 4 Follow-up ε, παρακολούθηση των συζητήσεων για το ψήφισμα για το TTIP. Θα θυμάστε ότι είχε γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στο σχέδιο γνωμοδότησής μου ως εισηγητή για το θέμα αυτό της Ατλαντικής Εμπορικής ε, Συμφωνίας. Έγινε μια συμφωνία μεταξύ σκιωδών Σήμερα είναι μια μέρα αφιερωμένη λίγο πολύ στην, στο TTIP. Ξέρετε ότι το απόγευμα θα έχουμε συζήτηση με την Επιτροπό Μάλμστρομ και θα γίνει μετά μια μίνι ακρόαση για το θέμα αυτό της συμφωνίας TTIP. Στην τελευταία συζήτηση έγινε έντονη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των σκιωδών για την έκθεση αυτή. και δεν μπορέσαμε τελικά να ακούσουμε όλους τους συναδέλφους που ήθελαν να πάρουν το λόγο. Ως εκ τούτου αποφασίσαμε να γίνει μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων εδώ σήμερα. Με μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε μια μισή ώρα στη διάθεσή μας για τη συζήτηση αυτή. και νομίζω ότι στη τελευταία συνεδρίαση παρουσίασα σε βάθος τα στοιχεία της έκθεσης. Οι σκιώδες εισηγητές, όπως σας είπα, πήραν το λόγο. Δεν θέλω να επαναλάβω λοιπόν αυτά που κάναμε την προηγούμενη φορά. Δεν θέλω να μιλήσω εγώ, θέλω να ακούσω τα δικά σας σχόλια. Και φυσικά όπως σας υποσχεθήκαμε την προηγούμενη φορά θα πάρουμε και θα συνεχίσουμε με τον κατάλογο αγορητών της προηγούμενης φοράς και μετά φυσικά θα ακολουθήσει η ανεκτή συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας. τα άτομα που ήταν στην προηγούμενο κατάλογο μελητών. Απόν, απόν, απόν, απόν. Και η κυρία Αρένα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πράγματι δύσκολο να συνεχίσει κανείς μια συζήτηση μετά από μερικών εβδομάδων διακοπή. Φαντάζομαι όμως ότι το θέμα TTIP θα παραμείνει στη μέση διάταξη πολύ καιρό. Με βάση αυτά που είπατε τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα γιατί είναι θετικά και επικοδομητικά σημεία για τη διαπραγμάτευση, ισορροπημένα και εγώ και η συνάδελφος Ζουντ την προηγούμενη φορά παρουσιάσαμε ορισμένες τροπολογίες και ομαδοποιήσεις τροπολογιών. Δεν θα σας εκπλήξει ότι η ομάδα μας είναι πολύ ευαίσθητη στο θέμα των δημοσίων υπηρεσιών και έγινε λόγος για θετικό και αρνητικό κατάλογο και το θέμα του αρνητικού καταλόγου μας θέτει πρόβλημα ιδιαίτερα για την προστασία των δημοσίων υπηρεσιών και εκεί βέβαια θα κάνουμε εναλλακτικές προτάσεις. Επίσης το θέμα του ISDS είναι θέμα επί του οποίου θα καταθέσει τροπολογίες η ομάδα μας και υπάρχουν και μερικά ακόμη σημεία ή θέματα που είναι συζητήσιμα για μας από τις προτάσεις σας γνωρίζοντας όμως ότι πρόκειται για επικοδομητική θέση ως προς το μέλλον των διαπραγματεύσεων αυτών. Είναι σημαντικό η Κομισιόν να ακούσει τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Δεν θα θέλαμε κατά το τέλος των συζητήσεων αυτών που κρατάνε τόσο καιρό να καταλήξει το κοινοβούλιο να αναγκαστεί να πει μόνο ναι ή όχι χωρίς να έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που διαθέτουμε εδώ στο Κοινοβούλιο για να περάσουμε όλα τα μηνύματα που θέλουμε στην Κομισιόν στους διαπραγματευτές ώστε με το άμα το πέρα τίτης να καταλήξουμε σε κάτι επικοδομητικό και ή δυνατόν αποδεκτό. Ευχαριστούμε πολύ και μερσή. Αν δεν είναι εδώ, Φλωρέντσα δεν είναι εδώ, ο κύριος Τσικάου όμως. Κύριε Τσικάου θέλατε να όχι, δεν. Ναι. Α, δεν, δεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι η πρότασή σας είναι σε αρχικό επίπεδο ένα αλλά μια καλή πρόταση. Είπαν όμως αρκετοί συναδέλφοι και την προηγούμενη φορά ότι έχει ανάγκη η πρόταση από κάποια επιπλέον στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να περιοριστώ στο να θέσω κάποια σημεία τα οποία είναι τεχνικού περισσότερο παρά πολιτικού χαρακτήρα. Σε επίπεδο πολιτικό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στα πλαίσια της αναζήτησης ε, μιας κάποιας ευκαιρίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρξει δηλαδή η μέγιστη δυνατή ε, δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις. Τώρα στο σημείο Α. Ε, αναφερόμενοι στα θέματα της εκ νέου ε, εκβιομηχάνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει θα έλεγα μια έλλειψη αναφορά συγκεκριμένα στον τομέα των υπηρεσιών. Ε, άνω του 35% ε, ε, ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και η διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας είναι πολύτιμο στοιχείο. Λοιπόν, στο γάμα 12 υπάρχει μια αναφορά θα έλεγα πιο συγκεκριμένη για τα θέματα της γεωργίας. Η γεωργία όπως γνωρίζετε είναι σημαντικό συστατικό των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του TTIP. Ε, συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσει να βρει λύσεις ε, για την ε, πρόσβαση των προϊόντων μας στην Αμερικανική αγορά καταργώντας τα μη δασμολογικά εμπόδια. Ένα άλλο τομέα είναι το να ληφθούν υπόψη τα διάφορα επίπεδα αλλαγών στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες εγγυήσει ε, για τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε ε, δημόσιες προμήθειες αμερικανικές. Νομίζω ότι έχουμε το παράδειγμα με τον Καναδά εδώ, τη συμφωνία με τον Καναδά που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Θα ήθελα να περιοριστώ σε αυτά λέγοντας ότι στα πλαίσια και των προσπαθειών του ISDS ε, νομίζω ότι μας είπε και ο Ιάπων πρέσβης τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το παγκόσμιο σύστημα ε, γίνεται μια συζήτηση για την δυνατότητα αυτή έτσι ώστε τα ISDS να είναι κάτι το θετικό, να είναι κάτι το οποίο ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας δικαίου και ταυτόχρονα να διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών. γιατί πολλές φορές οι επενδυτές βιώνουν τις νομικές ρυθμίσεις που τους αφορούν όχι σαν μια απλή εθνική νομική διευθέτηση, αλλά σαν κάτι το οποίο λειτουργεί συστηματικά εις βάρος των οικονομικών του συμφερόντων. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Λάγκε. Λείπει και ο κύριος Προύστ. Αλλά είναι εδώ ο επόμενος ο μιλητής, ο κύριος Φιέλνερ. Είναι πολύ καλή η έκθεσή σας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε πια να δημιουργούμε νέες κόκκινες γραμμές. Είχαμε μια έκθεση, υπενθυμίσαμε την άποψη του Κοινοβουλίου. Έχουμε την εντολή του Συμβουλίου. Δεν θα πρέπει λοιπόν εμείς να δημιουργούμε μια δεύτερη και μια τρίτη εντολή ανάλογα με τη συγκυρία. Διερωτώμε λοιπόν για το πώς θα αντιδρούσαμε εμείς σαν το Αμερικανικό Κογκρέσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων άρχιζε να παίρνει άλλες αποφάσεις μετακινώντας το τέρμα κάθε φορά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των ε, συζητήσεων ακούστηκαν ε, πολλά για το ε, ISDS. Είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε περισσότερο σήμερα το απόγευμα αυτά, υπενθυμίζω, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα από τα σημεία στα οποία Αυτά τα οποία λέτε κύριε Πρόεδρε δεν μου φαίνονται πάρα πολύ σωστά. Λέτε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο ίσως και να μην χρειάζεται. Ε, ένας άλλος ε, γερμανός σοσιαλδημοκράτης, ο Ζίγμα Γκάμπριελ, έχει πει ότι χρειαζόμαστε τα ISDS διότι θα προστατεύσουν τις επενδύσεις της νέας γενεάς. Είναι μια ευκαιρία τα ISDS έτσι ώστε να ορίσουμε υψηλότατα επίπεδα προστασίας των επενδύσεων παγκοσμίω. Και πρέπει να ακούσουμε το τι λέει ο Γερμανός αυτός σοσιαλδημοκράτης. Τώρα το λέω εγώ, εγώ αυτό, ακούγεται περίεργο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στο κομματικό έγγραφο της, του S5 στην Γερμανία και έχει πολύ ενδιαφέρον. Προσπάθησα να καταλάβω ακριβώς ποια είναι η θέση της σοσιαλιστικής ομάδας, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω το σύνολο των προτάσεων, αλλά λέτε ότι δεν θέλετε το ISDS, αλλά στο τέλος ε, λέτε ότι πρέπει να μεταρρυθμιστεί το ISDS και αν μεταρρυθμιστεί μπορεί να είναι ανεκτό. Νομίζω ότι δεν είναι κακή η θέση σας αυτή, ελπίζω να είναι τελικά η θέση του Κοινοβουλίου. Νομίζω επίσης ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της συζήτησης ε, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια θα πρέπει να λειτουργούν ή με το αν θα πρέπει να έχουμε δικαστήρια. Αντί να συζητήσουμε δηλαδή το περιεχόμενο του είδους της προστασίας την οποία θέλουμε τα δικαστήρια να παρέχουν, εμείς συζητάμε για το αν θα έχουμε ή όχι δικαστήρια. Νομίζω ότι εμείς σαν νομοθέτες θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας ε, όχι στα δικαστήρια αλλά στους νόμους και αυτό προσπαθώ να αποκαταστήσω με τις δικές μου τροπολογίες. Τι είναι σαν παράδειγμα δίκαιη μεταχείριση, ισότιμη μεταχείριση. Ναι. Ε, τι θα πει ε, έμεση, έμεση απαλωτρίωση τι ακριβώς ε, χρειαζόμαστε διαφορετικά επίπεδα προστασίας για διαφορετικού τύπου επενδύσεις. Νομίζω ότι αυτές είναι λεπτομέρειες οι οποίες ε, παρουσιάζουν ενδιαφέρον και μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτές αν ξεπεράσουμε τα υπαρξιακά ερωτήματα του στυλ θέλουμε δικαστήρια ή δεν θέλουμε δικαστήρια. Δυστυχώς λοιπόν κάποιες από τις προτάσεις σας δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Λέτε σαν παράδειγμα ότι δεν θέλετε προστασία, θέλετε ε, ε, προστασία μόνο για τις επενδύσεις μετά από την εγκατάσταση του επενδυτή στη χώρα. Ε, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η άποψη της σοσιαλιστικής ομάδας γιατί αν αυτή ήταν η άποψη τότε θα ήταν σωστό να κάνει κανείς διακρίσεις, αυτή τη στιγμή έχει πάρει μία επένδυση. Να πούμε ότι εμείς θέλουμε επενδύσεις σαν παράδειγμα μόνο από αμερικανικές επιχειρήσεις. Και αυτό είναι καλό γιατί ποτέ δεν θα έχετε την δυνατότητα να εγκατασταθείτε πλήρως και να αποκτήσετε έδρα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτά είναι λεπτομέρειες που δεν βλέπω γενικότερα στην εντολή την οποία έχουμε. Ένας άλλος τομέας είναι οι υπηρεσίες και η κυρία Ρενά αναφέρθηκε σε αυτές. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι όχι να φτιάξουμε ένα κατάλογο θετικό ή αρνητικό, αλλά θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να μην αποκλείουμε νέες υπηρεσίες, διότι ο τομέας των υπηρεσιών, ιδιαίτερα το ψηφιακό κομμάτι, μας δίνει συνεχώς νέα προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να περιορίσουμε το εύρος αυτής της ρύθμισης, γιατί ε, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις νέες υπηρεσίες. Δυστυχώς στα πλαίσια του TTIP ε, φοβόμαστε ε, για το τι μπορούμε, σε τι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς. Ας διευκρινίσουμε εμείς πρώτα το σε ποιους τομείς θέλουμε να συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς. Και φυσικά ε, τα θέματα της ροής των δεδομένων και γενικότερα ο ψηφιακός κόσμος είναι θέματα τα οποία άπτονται φυσικά και της ψηφιακής οικονομίας, αλλά όχι μόνο και της βιομηχανίας και των ε, χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Λοιπόν, ε, δεν μπορούμε να δεσμευθούμε αν ε, σαν παράδειγμα λέτε δεν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις νομοθετικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να περιορίζουμε τις φιλοδοξίες μας και δεν πρέπει να λέτε ότι δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις επειδή υπάρχει μια νομοθετική διαδικασία εν εξελίξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα είναι ιδιαίτερος δεσμευτικό. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα να ξεκινήσουμε με τον νέο κατάλογο ομιλητών. Το λόγο έχει ο κ. Βαλέσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική σας έκθεση. Επειδή πρόκειται να είναι μία από τις τελευταίες παρεμβάσεις, θα ήθελα να είμαι σύντομο. Καταλαβαίνω και χαίρομαι τις διατυπώσεις για το φυσικό αέριο και τις εξαγωγές από, το, από τις ΣΥΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η διατύπωση και μάλιστα σκοπεύω να καταθέσω σχετική τροπολογία. Να θέσω δύο σημεία. Καταρχάς, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ε, διατύπωση και να ξεκαθαρίσουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι η άρνηση των ΗΠΑ για να καταργήσει οποιασδήποτε φραγμού στην εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας κάνει πάρα πολύ δύσκολη την αποδοχή της πτυχής αυτής. Και κατά δεύτερον, οι σημαντικές εξαγωγές υδρογονοθράκων από τις ΗΠΑ πιστεύω ότι θα πρέπει να συνοδεύονται από μια προστασία του δικού μας κλάδου, από μια μεγάλη περίοδο εξαίρεσης που θα ξεκινήσει όταν θα υπάρξει ροή πλέον ε, φυσικού αερίου και πετρελίου από τη ΣΥΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το πακέτο κινητικότητας. Πιστεύω ότι δεν έχουμε βρει ακόμα τη σωστή διατύπωση γιατί το πακέτο κινητικότητας είναι ύψης της σημασίας και η διευκόλυνση των θεωρήσεων για τις ε, Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για την εκμετάλλευση, την αξιοποίηση, την πλήρη αξιοποίηση της συμφωνίας TTIP. Θα καταθέσω λοιπόν τις σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος, ο κ. Ζαντό. Ευχαριστώ, Μπέρντ. Πράγματι δεν θα επαναλάβουμε όλα όσα έχουν ξαναϋποθεί στο προηγούμενο πρώτο τμήμα της συζήτησης. Απλώς μερικά σχόλια για την συνεργασία, δικανονιστική συνεργασία Πρέπει φυσικά να ενδυναμωθεί η αποτίμηση, αξιολόγηση, αντικτύπου κτλ. επί των καταναλωτών και τέτοια. Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι μια απλή υπενθύμηση των ευθυνών που έχουν οι υπεύθυνοι γιατί προβλέπονται όλες αυτές οι αξιολογήσεις. Το ενδιαφέρον όμως θα ήταν εφόσον το θέμα αρχίζει να συζητιέται ευρύτερα θα ήταν να δούμε τι επιπτώσεις έχει, πώς να το πούνε, το chill effect, δεν ξέρω πώς να το πω, κάποιο είδους σχετικό πάγωμα των νομοθετικών διαδικασιών γιατί δεν ξέρουμε αν πρόκειται για πραγματική συνεργασία εκ των προτέρων ή αν μόνιμα θα τα εξετάζουμε όλα νομοθετικά μόνο υπό το πρίσμα των επενδύσεων και του εμπορίου και των ανταλλαγών, συναλλαγών. να το δούμε και αυτό το θέμα του chill effect δηλαδή. Έπειτα τα χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, δυστυχώς στο TTIP αυτό δεν προβλέπεται ούτε συνεργασία, ούτε δυνάμωση, ούτε περισσότερη εποπτεία και συνεργασία μεταξύ των εποπτών από Αμερική και Ευρώπη για να αποφευθούν καταστροφές όπως το 2008 και μία σύγκληση των κανόνων εδώ θα κατέληγε στη δημιουργία ενός πολύ βαρύτερου κινδύνου, σοβαρότερου κινδύνου ίσως λιγότερο στο γενικότερο σύστημα αλλά μεγαλύτερο σε ορισμένες χώρες και γενικότερα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα γιατί όλοι οι εμπειρογνώμονες λένε ότι τα μαθήματα του 8 δεν τα πήραμε υπόψη μας και ότι άρα υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί η ευαλωτότης του συστήματος. Για το SDS η θέση του εισηγητή είναι η θέση του μέλλοντος. Κοιτάξτε πώς εξελίσσεται η συζήτηση στα ΣΥΠΑ. Και στο Κογκρέσο ακούγονται πράγματα από επιφανής νομομαθής ότι το ESDS είναι σύστημα που δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και υπάρχουν και think tanks και ιδρύματα, Ινστιτούτα που δεν είναι από τα πιο προοδευτικά που παραδέχονται ότι όπως το Ίδρυμα Αγρόπα Νόστρα και του Ζακ Ντελόρ και τα λοιπά που παραδέχονται λέγω ότι δεν είναι σίγουρο καθόλου ότι όλα αυτά είναι τα δέοντα. Δεν θέλω να κάνω σαν τον Φιέλνερ ένα είδου ταλμουδικής εξήγηση ε, της ε, σοσιαλιστικής θέσης για το ΙΕΣΔΑΕΣ, αλλά να αναφερθώ συγκεκριμένα στην ψηφιακή οικονομία που δείχνει πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημα του ESDS. Τι είναι η ψηφιακή οικονομία. Είναι κεφαλαιοποίηση κατά 85% για τους Αμερικανούς, κατά 2% για τους Ευρωπαίους. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι η Γερμανία θα είχε κάποτε πρόβλημα με το σύστημα Uber. Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και γι' αυτό οι επιχειρήσεις, οι ψηφιακές επιχειρήσεις αντιτίθενται στο ESDS. Γιατί θα εμποδίζει ό,τι μέτρα και να ληφθούν την ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί στην Ευρώπη. Ούτε για την προστασία των δεδομένων, ούτε για τα φορολογικά δεν θα ισχύει. Επομένως, το παράδειγμα αυτό της ψηφιακής οικονομίας είναι τέλειο παράδειγμα της αποτυχίας του ESDS. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κεκέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Προσωπικά είμαι υπέρ της σύμφωνίας του TTIP και θα πρέπει να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Αλλά η ουσία είναι ότι θέλουμε μια ανταγωνιστική Ευρώπη. Αν δεν διαπραγματευτούμε το TTIP θα μας θέσει σε μειονεκτική θέση αυτό στο μέλλον σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο εμπόριο. Συμφωνώ αρκετό, αρκετά με αυτά που είπε ο κύριος Φιέλνερ για τα όρια που υπάρχουν. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν κάποιες ε, γραμμές που δεν θα ξεπεραστούν σε κάποια θέματα στη γεωργία. Δεν έχει νόημα να λέμε ότι δεν θέλουμε να συμπεριληφθεί η γεωργία στο TTIP. Θέλουμε και πρέπει. για τις ε, σχετικές στασιστικά μηχανήματα, για παράδειγμα. Προφανώς ε, αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή, γιατί δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε αυτά. Πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να δεχτούμε και τι δεν μπορούμε να δεχτούμε. Αλλά γενικότερα, όπως είπε ο κύριος ε, Φιέλνερ, σε ό,τι αφορά το ψηφιακό τομέα που αλλάζει κάθε ημέρα και αυτό θα συνεχιστεί, αυτό σημαίνει καινοτομία. Όσα μας είπε λοιπόν ο κύριος Χέλνερ για να υπάρχει μια προετοιμασία για το μέλλον, είναι πολύ σημαντικό. Και προφανώς η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι η βασική πρωτοπόρη του μέλλοντος. Δεν θέλουμε αυτό να το διακυβεύσουμε για το ISTS. Σημαντικό και αυτό. Στα πλαίσια του TTIP. Έχω μιλήσει με τους εκπροσώπους ε, του εμπορικού κλάδου στην χώρα μου και ανησυχούν ιδιαίτερως. Αλλά πιστεύω ότι οι εξελίξεις ε, με τη συμφωνία ΣΥΤΑ δείχνουν το πώς μπορούμε να εξελίξουμε το STS και να το καταστήσουμε λειτουργικό. αυτή τη γραμμή θα πρέπει να ακολουθήσουμε και όχι να λέμε ότι δεν το θέλουμε το σύστημα αυτό καθόλου. Νομίζω λοιπόν ότι έχει γίνει καλή δουλειά, το σημειώνουμε πρόοδο, περνάνε οι θέσεις μας, αλλά να μην φοβόμαστε γιατί σε τελική ανάλυση θα ψηφιστούν αυτά. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ναι ή όχι. Ας συζητήσουμε λοιπόν και σε τελική ανάλυση πάντα μπορούμε να αποφασίσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντινγκ έχει το λόγο. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για τη σημαντική δουλειά που κάνατε ως εισηγητής για την έκθεση αυτή. Να σχολιάσω λίγα μόνο στοιχεία τα οποία με απασχολούν ιδιαίτερως. Για τις υπηρεσίες καταρχάς. Όπου νομίζω ότι η έκθεση μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Τηλεπικοινωνίες σε ό,τι αφορά το, το κομμάτι της ε, προσβασιμότητας στην αγορά. Ο δικέ μας απασχολεί το θέμα αυτό και θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να έχουν πρόσβαση οι Ευρωπαίοι προμηθευτέ παροχή στην Αμερικανική αγορά. Γιατί είναι απαγορευτικά τα πράγματα σήμερα. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, θεωρώ ότι πρέπει να πούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η προστασία των δεδομένων και η τωρινή και η μελλοντική θα πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστή. Και δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε δέσμευση, να λάβουμε οποιαδήποτε δέσμευση για με την κατάσταση της επεξεργασίας των δεδομένων εφόσον δεν υπάρχει επίλυση των θεμάτων της ε, ρύθμισης, της κανονιστικής διαδικασίας μεταξύ Ευρώπης και ΕΠΑ. Έχει υπογραμμιστεί ότι το TTIP θα πρέπει να αποτελέσει φραγμό για την ανάπτυξη της ψηφιακής ατζέντας της Ευρώπης, αλλά το TTIP θα πρέπει να μας επιτρέψει να αναπτύξουμε ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού μια κοινή ψηφιακή οικονομία προκειμένου να υπάρχει αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά και ίση όρη. Εδώ λοιπόν πολλά θα πρέπει να γίνουν ακόμα. Ξέρω ότι το συζητήσαμε το ISDS και θα το συζητήσουμε και πιο επισταμένος. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι, κυρία εισηγητά, η έκθεσή σας πάει πολύ υπερβολικά μακριά. Ξεπερνάει κάποια όρια. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένας μηχανισμός ο οποίος θα εξασφαλίσει την προστασία των επενδύσεων. Δεν πιστεύω δε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια... Η λύση μπορεί να είναι μια επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών, γιατί αυτό ενδεχομένω ε, να οδηγήσει στην ε, μη τήρηση της δημοκρατικής ε, νομοθεσίας. Ούτε νομίζω ότι είναι κατάλληλος ο τρέχον μηχανισμός δεν τηρεί βασικές δικαστικές αρχές, ούτε εξαρτησία βλέπουμε, ούτε την αμεροληψία των δικαστών που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας μας. Ούτε υπάρχει η συνοχή, η ομοιογένεια και η προβλεψιμότητα των αποφάσεων. Ξέρω ότι θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε τη μεταρρύθμιση ενός συστήματος το οποίο περιλαμβάνεται σε 14.000 διμερείς συμφωνίες ήδη και η μεταρρύθμιση γίνεται και στην συμφωνία ΣΥΤΑ θα αρκέσει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ προσωπικά πιστεύω επειδή δεν αρκεί να επιλύσουμε το πρόβλημα σε αντιμερές επίπεδο με τη ΣΥΠΑ, θα πρέπει να επιλύσουμε το θέμα αυτό των 1.400 διορθώνει ο Μιλήτρια, συμφωνιών σε ό,τι αφορά τους δικαστές που ορίζονται για μια συγκεκριμένη περίοδο για την εξέταση των διεθνών προτύπων. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο για να επιλύσουμε τα θέματα που προκύπτουν και μεταξύ των πολιτικών ομάδων για να συμφωνήσουμε δηλαδή για μια κοινή λύση. Δεν θα επισέλθω τι λεπτομέρειε. Θα πω μια τελευταία κουβέντα, Πρόεδρε. Λαμβάνοντα υπόψη τι πρόσφατε εξελίξει στην Ευρώπη για το TTIP, πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια έκθεση. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε με σαφήνεια τι συστάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό λοιπόν θα καλέσω τα κρατημέλη να καταθέσουν συμβιβαστικέ τροπολογίες, γιατί θα πρέπει στη σημερινή κατάσταση να έχουμε μια ισχυρή ενιαία θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί πιστεύω ότι στη τελική ανάλυση, αν λάβουμε τις σωστές αποφάσεις, αν ε, σχεδιάσουμε με τον σωστό τρόπο την συμφωνία TTIP θα έχει σημαντικές ωφέλειες και πλεονεκτήματα και για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Κύριος Στήρ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω τα, την κρατική γλώσσα. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον προηγούμενο συνάδελφο και να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που κάνατε για να προετοιμάσετε αυτή την συμφωνία. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω και για, την, για το σωστό πνεύμα ε, συνεργασίας το οποίο επιδείξατε. Να ευχαριστήσω επίσης και την Επιτροπή Ανάπτυξης η οποία έχει ε, ακολουθήσει σωστή γραμμή και νομίζω ε, παράλληλα ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ανοίγονται νέες ευκαιρίες στον τομέα της ανάπτυξης ε, από την ε, συμφωνία αυτή, την ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τον μηχανισμό ε, επίλυσης διαφορών ή μηχανισμό διαιτησίας αν θέλετε. Προέρχομαι από μια νέα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κροατία ένας τέτοιος μηχανισμός ο οποίος ε, ε, θα ξεπερνά τις εθνικές ε, δικαιοδοσίες είναι κάτι το θετικό νομίζω γιατί ενισχύεται η εικόνα η οποία πρέπει να ισχύει για την προστασία των ξένων επενδυτών. Θα πρέπει δηλαδή ε, να κατανοούν οι επενδυτές ότι την χάνουν των ιδίων εγγυήσεων είτε σε μια μικρή χώρα όπως είναι η Κροατία είτε σε μια μεγαλύτερη και παλιότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια σημαντική πλευρά η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το να πιστέψει κανείς ότι δεν χρειάζεται κανένας έναν μηχανισμό όπως το ISDS ε, είναι αρνητικό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόβλημα όταν παίρνει το λόγο κανείς ε, στο τέλος μιας συζήτησης ε, είναι ότι έχουν υποθεί όλα τα πιο σημαντικά πράγματα και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την έκτασή σας και ουσιαστικά τώρα κάνουμε απλά μία ενημέρωση. Και από όλες ε, τις τοποθετήσεις σας, από όλες τις τροπολογίες που θα κατατεθούν, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ομοιογενές σύνολο. Καταρχάς να πω ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρη κατά πόσον στην παρούσα χρονική φάση χρειαζόμαστε κατεπηγόντως μία έκθεση αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια συνεκτική έκθεση, την οποία την υποστηρίζει η πλειοψηφία. Αν δεν υπάρχει αυτή η έκθεση, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια συνένεση, είναι σημαντικό αυτό. Αυτό που θα ήταν καλύτερο θα ήταν να έχουμε μια συνεκτική έκθεση, το οποίο να έχει ευρεία υποστήριξη. Πρώτη λοιπόν παρατηρήση που έχω να κάνω. Το έχω επισημάνει και στο παρελθόν στις συζητήσεις μας. Διαβάζοντα, διαβάζοντας την έκθεση, δεν μου δίνει την εντύπωση ότι μιλάμε και για άλλους. Πιο πολύ ότι μιλάμε για την επιβέβαιση των δικών μας προτύπων. Αυτό δεν είπατε. ένα αμφιβόλο. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο, όπως είπε και ο συνάδελφος Ζαντό. Ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις για τις συνέπειες του ευρωπαϊκού μοντέλου. Αλλά υπάρχει το ευρωπαϊκό μοντέλο. Εξακολουθώ να έχω την αίσθηση λοιπόν ότι κάποιες διατυπώσεις μπορούν να είναι πιο θετικές. Με την κοινή λοιπόν έκθεση από πλευράς του Κοινοβουλίου δεν θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε κατά βάση δεν θέλουμε την συμφωνία, εντάξει τη συζητάμε μεν αλλά κατά βάση είμαστε κατά. Αυτό ως γενικό σχόλιο. Γιατί υπάρχει πάντα ένας ψυχολογικός ε, παράγοντας, μια συναισθηματική φόρτιση, η οποία πάντα παίζει το ρόλο της. Και πιο συγκεκριμένα. Δεν πρόκειται να συνεχίσω να συζητώ τον όρο ISDS από εδώ και πέρα. Αλλά πιστεύω ότι μια προστασία των επενδυτών με μια αναθεωρημένη μορφή είναι κάτι το εντελώς απαραίτητο. Και ότι ως κοινοβούλιο μπορούμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία αυτή για να ορίσουμε Ποιε είναι οι δυνατότητε που θεωρούμε ότι υπάρχουν. Σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουμε με την Επίτροπο. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να διαμορφώσουμε μία άποψη. Ίσως ένα ΣΥΤΑ συν να αποτελέσει ένα μοντέλο. Ίσως να υπάρχουν και άλλα μοντέλα. Αλλά σίγουρα όχι υπό την ε, σημερινή μορφή. Θέλουμε μία αναθεωρημένη μορφή και θα πρέπει να τα συγκεκριμενοποιήσουμε όλα αυτά. Κατά δεύτερον, για τις υπηρεσίες. Νομίζω ότι τα ακούσαμε ήδη. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα πρέπει να αλλάξει η προσέγγιση μας σε σχέση με την προσέγγιση που ακολουθήσαμε στο ΣΥΤΑ. Εγώ είμαι υπέρ ενός αρνητικού καταλόγου. Να σας πω και γιατί. Γιατί πολλά από αυτά που συζητάμε βασίζονται σε αυτά που ισχύουν σήμερα, το 2015. Μία κατάσταση ίσως που γνωρίσαμε, με την οποία μεγαλώσαμε, με μια οικονομία η οποία ήδη υφίσταται. Αυτό που θέλουμε να οικοδομήσουμε είναι κάτι για το μέλλον. Για την επόμενη περίοδο που θα μας χρησιμεύσει μεσοπρόθεσμα και η ταχύτητα των εξελίξεων στην οικονομία, στην βιομηχανία. Είναι κάτι το αντιαφισβήτητο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν στο μέλλον. Αν κάνουμε ένα θετικό λοιπόν κατάλογο σήμερα, δεν λαμβάνουμε υπόψη το τι θα ισχύει ενδεχομένως 15-20 χρόνια. Πραγματικά λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την προσέγγιση που ακολουθήθηκε στη Συμφωνία ΣΥΤΑ. Χρειαζόμαστε δεσμευτικούς κανόνες για βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, δεν είμαι καθόλου βέβαιη αν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξαναγκάσουμε τη ΣΥΠΑ να επικυρώσουν οποιασδήποτε διεθνείς συμβάσεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε αυτά που ισχύουν εδώ. Αν θέλουμε το σύστημα μας, αυτό το αποκαλέσουμε έτσι, να γίνει σεβαστό, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία αμοιβαιότητα. Να πούμε κι εμείς ότι και εσείς ε, στη ΣΥΠΑ μπορεί να ακολουθήσετε το δικό σας σύστημα, το σεβόμαστε. Και ενδεχομένως στο μέλλον να χρειαστεί να ψάξουμε μεγαλύτερη συμβατότητα. Θα προσπαθήσουμε από πλευρά της ομάδας μας να καταθέσουμε συνεκτικές, ε, εναρμονισμένες τροπολογίες. και σίγουρα προσβλέπω στις μελλοντικές ε, εργασίες μας και είμαι πεπισμένη ότι θα πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πρόεδρος, κυρία Μπικίν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρό μας για μια πολύ καλή έκθεση έδειξε θάρρος, στις, επέμεινε στις θέσεις του και στον τομέα του ISDS. και δεν δέχθηκε τις πιέσεις ε, έτσι ώστε να μην συμπεριληφθεί το ISDS στη συγκεκριμένη πρόταση, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε βέβαια αλλά έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα για το θέμα της διατησίας ή της δικαστικής προστασίας. Ε, δεν μπορούμε εμείς να τα παραπέμψουμε όλα σε ένα διεθνές ιδιωτικό δικαστήριο, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να χάσουμε και ε, μια τόσο μεγάλη ευκαιρία για δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε εμείς να εκχωρήσουμε τη δικαιοδοσία μας σε ένα, ε, ε, σε ένα διεθνές δικαστήριο υψηλού επίπεδου και δεν μπορούμε επίσης να μειώσουμε και την ποιότητα των προϊόντων τα οποία καταναλώνουμε στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνετε στην πρότασή σας κύριε ε, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα όμως να εμείνετε λίγο περισσότερο στην βασική αρχή της πρόληψης. Εφόσον υπάρξει μια συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες, θα θέλαμε να μας ε, δηλώσουν ότι ανοίγουν πλήρως τις δημόσιες προμήθειές τους, ε, ενώ οι δικές μας είναι ήδη ανοιχτές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ να τεθεί και το θέμα και της αναγνώρισης των επαγγελματικών ικανοτήτων, πτυχίων κτλ. Ε, είναι πολλές οι κοινοβουλευτικές επιτροπές οι οποίες γνωμοδοτούν γύρω από το θέμα αυτό. Οι περισσότερες έχουν εκφράσει τη θέση τους για το TTIP. Σε πολλές ε, επιτροπές υπήρξε συμφωνία στα περίπλοκα πράγματι θέματα τα οποία θέτει η συμφωνία αυτή. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να αγνοήσουμε τον κόπο των συναδέλφων. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις για την μέθοδο εργασίας την οποία θα ακολουθήσουμε από τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πρόεδρε και εισηγητά. Είναι πολύ σημαντικό να μην παραλείψουμε τίποτε από αυτά που μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε στην αρχή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ταυτίσουμε ως θετικό να μην θεωρείται μόνο ένα κατάλογος κόκκινων γραμμών αρνητικά δηλαδή, αλλά να δούμε και τι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να δείξουμε ότι αυτό θέλουμε, ότι έχουμε υψηλές προσδοκίες, ότι θέλουμε να πάρουμε αυτή την ευκαιρία υπέρ των πολιτών μας. Τώρα βέβαια είναι και αυτοί που δεν θέλουν τη διαπραγμάτευση, αλλά αυτούς τους παρακαλώ να μην υποβάλουν πολλές τροπολογίες, γιατί εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε κείμενο που να βοηθάει τη διαπραγμάτευση με, τις, με τα θετικά σημεία που θέλουμε, επί των οποίων θέλουμε να επιμείνουμε. Να μην τα παραλείψουμε λοιπόν αυτά. Να δηλώσουμε σαφώς τι θέλουμε ακριβώς από αυτήν. Όχι μόνο τι δεν θέλουμε αλλά και τι θέλουμε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα συνεχίσουμε την καλή συνεργασία για να πετύχουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για τους πολίτες μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Θέλω να θίξω δύο θέματα για το ISDS. Γιατί πιστεύω ότι το θέμα με το TTIP δεν είναι ότι δεν το χρειαζόμαστε. Αλλά ότι πρόκειται για πολύ προβληματικό τρόπο επίλυσης διαφορών και πολύ λαθεμένο. Η προφανής εναλλακτική επιλογή θα ήταν να επιλύονται οι διαφορές από εθνικά δικαστήρια. Άρα και για επενδυτές. Νομίζω ότι θα ήταν αρνητικό να υπάρχει ένα ειδικό δικαστήριο για τους επενδυτάς. Πρέπει να βασιστούμε στα τοπικά δικαστήρια και τοπικά δικαστικά συστήματα που υπάρχουν και στη ΣΥΠΑ και σε εμάς και έτσι μπορεί καμιά φορά οι επενδυτές να χάσουν και μια δίκη. Τώρα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η έκθεση συνδέει αυτό το θέμα με την σύγκληση σε υψηλότατο λέει επίπεδο Α, συμφωνώ βέβαια, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι στη ΣΥΠΑ εφαρμόζονται μειώσεις των προτύπων και των προδιαγραφών. Εμείς δεν δεχόμαστε, πρέπει να πούμε, τέτοιους περιορισμούς. Αυτό είναι το κυριότερο να υπάρξουν υψηλότερες προδιαγραφές αλλά επίσης να διασφαλιστεί ότι δεν θα μειώνονται και θα εφαρμόζονται αυτά οι προδιαγραφές. Έπειτα η έκθεση ζητάει για αξιολόγηση αντικτύπου για να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις και επί των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Και με αυτό συμφωνώ, αλλά Ήδη υπάρχει αυτό στην αξιολόγηση στο, στην, που έχει ήδη προβλεφθεί. Τι θα την κάνουμε όμως αυτή την πληροφόρηση. Να μην παραμείνει απλώς στα χαρτιά αλλά να είναι δεσμευτική να υπάρχει υποχρέωση. υποχρέωση. γιατί μπορούν να γίνουν πολλές αξιολογήσεις αλλά οι, τα συμπεράσματά τους δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε επικοδομητικά ούτε αλέως. Αυτές οι αξιολογήσεις λοιπόν καθεαυτές δεν μας βοηθάνε. Αυτά ήθελα να σας πω και σας κατευχαριστώ. Ο Χέλμουτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ είχα τη δυνατότητα να πάρω το λόγο ε, εκτεταμένα στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζουμε την γενικότερη κατεύθυνση της έκθεσης, γιατί κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα βασικά, κεντρικά ερωτήματα, τα οποία ανακύπτουν με το TTIP. Αλλά να αναφερθώ σε τρία-τέσσερα σημεία. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τρέχουσα χρονική στιγμή θα πρέπει να τοποθετηθεί. Γιατί πρόκειται για μια δημοκρατική άσκηση, ένα δημοκρατικό εγχείρημα. Ρωτήσατε κατά πόσον έχει νόημα, συνάδελφε, να τοποθετηθεί με αμφιλεγόμενο τρόπο ή ίσως με λιγότερο ξεκάθαρο τρόπο το Κοινοβούλιο. Όχι. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια έκφραση της δημόσιας συζήτησης, για ένα βασικό ζήτημα, για ένα ουσιώδες ζήτημα. Πρόκειται για μια συζήτηση πολλών μηνών όπου προσπαθούμε να προτιμήσουμε την ε, να σχηματίσουμε άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό αποτελεί τμήμα της προσπάθειας να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του δημοκρατικής ευθύνης. Έχει αυτό συνέπειες. Και εδώ θα επανέλθω σε αυτά που είπα και την πρώτη φορά. Το TTIP ε, για μια διατλαντική αγορά. Τίθεται λοιπόν το θέμα ποια κανονιστικά πρότυπα έχουμε, αυτή η αγορά ποιους κανόνες θα ακολουθήσει και πώς λειτουργεί η εσωτερική αγορά που υπάρχει μέχρι σήμερα σε σχέση με την ελεύθερη ζώνη εμπορίου της Βορειοαμερικής. Και αν θέλουμε να σχηματίσουμε μια κοινή αγορά από τις πολύ διαφορετικές αυτές ελεύθερες ζώνες, θα πρέπει να το εξετάσουμε επισταμένο στο ζήτημα λοιπόν αυτό. Αυτό αφορά η συζήτηση. Για το ESDS θα μιλήσουμε σήμερα το απόγευμα. Μία παρατηρήση επιτρέψτε μου. Θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουμε να εγκαθιδρύουμε την ιδιωτική αυτή επίλυση διαφορών σε κοινωνικά ζητήματα. Αυτό ίσως να το χρειαζόμαστε στον 20ο αιώνα, όχι όμως στον 21ο. Και η κυρία Ρέντινγκ έθεσε ένα πολύ ενδιαφέροντα παράγοντα για το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν τα χρήματα πιστοτικά, τα οικονομικά δικαστήρια. Δεν χρειαζόμαστε, θεωρώ, να τα αποφασίσουμε θέματα τέτοια πριν αποφασίσουμε για το συνολικό θέμα του ESDS. Στις ε, πολλαπλές ε, διμερείς συμφωνίες που υπάρχει η ρήτρα ESDS έχει επανέλθει στην ημερήσια διάταξη και πιστεύω ότι ένα διεθνές ε, τέτοιο οικονομικό δικαστήριο το οποίο θα έπρεπε να επιλύει διαφορές, αλλά όχι βάσει ιδιωτικού δικαίου, θα μπορούσε να αποσελέσει τμήμα της λύσης. Δεν ξέρω χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση εδώ στο ΣΥΤΑ και στο ΤΙΤΙΠ και πιστεύω ότι αν κοιτάξουμε τις συζητήσεις που γίνονται στο Κογκρέσο γίνεται ακριβώς η ίδια ανταλλαγή απόψεων και πολλοί και εκεί αναρωτιούνται κατά πόσο χρειάζεται το ISDS. Τρίτον, μιλήσαμε για δεδομένα. να σας πω ότι υπάρχει ένα σχέδιο ενοποιημένου σχεδίου κειμένου για το θέμα αυτό, για τις τηλεπικοινωνίες. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτά όντως είναι απαραίτητα για την ροή δεδομένων και πιστεύω ότι χωρίς προστασία των δεδομένων, χωρίς σχετική συμφωνία για την προστασία των δεδομένων, Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Χρειαζόμαστε σαφή ρυθμίση και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την ε, υφιστάμενη οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Να επισημάνω και συνταν και οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις στην Βουλγαρία και στην Ολλανδία για τις εθνικές ε, νομοθεσίες οι οποίες ε, ακυρωθήκαν και στη Γερμανία υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση. Θα πρέπει να κάτσουμε θεωρώ να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με την προστασία των δεδομένων σε ό,τι αφορά και την μελλοντική συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Και αυτό γιατί τα δεδομένα είναι προϊόντα, προϊόντα εμπορεύσιμα, που τα εμπορεύονται. Ως εκ τούτου λοιπόν, πιστεύω ότι είναι καλό το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ένα τόσο βασικό ζήτημα και όλα όσα γίνονται και στις άλλες επιτροπές που συζητούν άλλες πτυχές του ζητήματος, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί δεν είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά θα έπρεπε και θα θέλαμε να είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να επηρεάσουμε την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεσή σας είναι γενικά μια καλή και ισορροπημένη έκθεση. Πρέπει όμως να ενισχυθεί ακόμα σε ορισμένα σημεία. Θα συμφωνήσω με ορισμένους προλαλήσαντες όπως την ΕΜΑ. Το θέμα είναι να δούμε τι μήνυμα θέλουμε να στείλουμε. Το μήνυμα είναι ότι υποστηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές ε, απλά πρέπει να υπογραμμίσουμε ποια είναι τα συμφέροντα τα οποία εμπλέκονται εδώ και με ποιο τρόπο επιθετικό ή αμυντικό δρούν τα συμφέροντα αυτά. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι το TIP είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να ενισχύσει την ενιαία αγορά να της επιτρέψει να αναπτυχθεί δεν θα επιλύσει όλα τα προβλήματά μας αλλά νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να το διευκρινίσουμε κάπως καλύτερα στην παρουσίασή σας. Θα σταθώ τώρα σε τρία επιμέρους στοιχεία, τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο την Επιτροπή ΙΝΚΟ. Λοιπόν, ο τομέας των υπηρεσιών ένα τρίτο περίπου του συνόλου του κύκλου εργασιών ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι κάτι που πρέπει να ενισχυθεί στην έκθεσή σας. Διαφωνώ με την πρότασή σας για τον λεγόμενο αρνητικό κατάλογο. Αντίθετα νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά στα πλαίσια της λεγόμενης θετικής λίστας, του θετικού καταλόγου, στα πλαίσια τώρα των κρατικών προμηθειών. Αυτό είναι βασικό θα έλεγα στοιχείο και εδώ οι διαπραγματευτές θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο έτσι ώστε να διασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε και σε επίπεδο ομοσπονδιακό αλλά και σε επίπεδο πολιτιακό. Νομίζω ότι θα πρέπει να το διευκρινίσετε στην έκθεσή σας. Τώρα το, ε, η διακανονιστική συνεργασία και τα κοινά επίπεδα προστασίας. Νομίζω ότι εδώ βρίσκεται η καρδιά των διαπραγματεύσεων. Αν έχουμε μπορούμε να έχουμε κοινά επίπεδα προστασίας ε, ή αν μπορούμε τουλάχιστον να συνεργαζόμεθα πριν καθορίσουμε τα επίπεδα συνεργασίας και προστασίας τότε θα αποφύγουμε πάρα πολλές διαφορές ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν η σύγκληση η διακανονιστική που θα ωφελήσει τις μικρομεσαίες να είναι στόχος. Ε, σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τα ISDS. Θα συμφωνήσω με την κυρία Ρέντινγκ εδώ. Η διατύπωση η ισχύουσα είναι η χειρότερη επιλογή. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε το TIP για να μεταρρυθμίσουμε τα ISDS τότε θα μείνουμε πραγματικά ε, ουραγοί. Το ISDS είναι κάτι το οποίο χρειάζονται οι διεθνείς επιχειρήσεις ε, γιατί δεν μπορούν ε, οι διεθνείς διαιτησίες να αποφασίζονται με βάση τις πολιτιακές σαν παράδειγμα ή περιφερειακές αμερικανικές ρυθμίσεις. Το θέμα λοιπόν του δικαστηρίου στα πλαίσια του ISDS είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε. Αλλά απαιτείται να υπάρχει ενός κάποιου τύπου μηχανισμός. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε με δεκτικό τρόπο το τι ε, ε, μέτρα μπορούμε να πάρουμε για να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε τον μηχανισμό αυτό το ISDS. Θα τα πούμε και με την κυρία Μάλστρομ. Σίλβα. Και μετά θα πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Σίλβα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους Θα ήθελα να πω ότι η έκθεσή σας είναι ε, μια πολύ ε, ισορροπημένη και θετική έκθεση και έρχεται σε μια πολύ εύθετη στιγμή των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι είναι επίκαιρη επίσης γιατί πρέπει να στείλουμε στους διαπραγματευτές ένα ξεκάθαρο και χρήσιμο μήνυμα για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν δύο σημεία στα οποία θα μου επιτρέψετε να επιμείνω. Είναι δύο σημεία τα οποία θα μπορούσαν με χρήσιμο τρόπο να συμπληρώσουν την συμφωνία. Το πρώτο αφορά την κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα, στον τομέα των εξαγωγών. Ε, επίσης είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει άμεσα φυσικά και τους επενδυτές. Θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε με ποιο τρόπο λειτουργεί ένα σύστημα διεθνών συναλλαγών. Υπάρχει επίσης το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων, ικανοτήτων, διπλωμάτων. Ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και στην παρούσα φάση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να ε, ορίσει τις θέσεις της καλύτερα όπως και η Αμερικανική. Έρχομαι τώρα στο κεφάλαιο της προστασίας των επενδυτών. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε μια συζήτηση εκ νέου, άλλωστε θα ακούσουμε την άποψη της κυρίας Μάλιστον το απόγευμα. Κατανοώ πλήρως όμως την παρατήρηση την οποία κάνατε, λέγοντας ότι έχουμε ανάγκη από ένα ευρύτατο κεφάλαιο γύρω από το θέμα της προστασίας των επενδύσεων. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης γενικότερα για τις μορφές διαιτησίας. Ανεξαρτήτως αν υπάρχει ε, μια προβλεπόμενη μορφή διαιτησίας ή δεν υπάρχει μια τέτοια πρόταση στην τελική μορφή της έκθεσης, πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου. Πρέπει να προστατεύσουμε ε, ε, τα συστήματα αυτά ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενός συστήματος διεκτησίας ή μη. Εάν υπάρχουν κάποιες καταχρήσεις, σαν παράδειγμα της έννοιας της έμεσης απαλωτρίωσης, τα θέματα αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν είτε σε ένα διαιτητικό δικαστήριο είτε σε ένα εθνικό ε, δικαστήριο. Ε, λοιπόν, εμείς ε, το θέμα αυτό ή πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε αφεαυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να μιλήσουμε για τη διαιτησία θεωρητικά. Πρέπει να μιλήσουμε για τα ωφέλη τα οποία μπορεί να έχει την επενδυτική δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε κάποιο περιθώριο εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. όχι πάνω από 15 λεπτά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είμαι σύντομος. Γιατί η συζήτηση ήταν πολύ θετική, την άκουσα με προσοχή και μερικά από αυτά που υπόθηκαν θα τα μεταφέρω στην Επίτροπο Μάνστρομ που όπως ξέρετε θα έρθει το απόγευμα για να σας μιλήσει. Επομένως δεν θα αναφερθώ για το θέμα της, ε, που θα συζητήσει το απόγευμα θα περιοριστώ σε μερικά σχολιάκια. Είναι προφανές ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό ψήφισμα και θα εγκριθεί σε πολύ σημαντική στιγμή αυτών των διαπραγματεύσεων. Επίσης είναι σαφές ότι η πολιτική συγκυρία στη ΣΥΠΑ έχει γίνει πιο δύσκολη από την τελευταία φορά που μιλήσαμε όπου κυριαρχούσε κάποια αισιοδοξία. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα από ό,τι νομίζαμε ως διαδικασία έγκρισης. Η ιδέα ότι μέχρι Απρίλιο-Μάιο θα έχουμε καταλήξει δεν είναι, δεν σταθή. Μετά το καλοκαίρι μάλλον. Would Πολλοί από εσά μιλήσατε για το θέμα των κοκκίνων γραμμών. Φυσικά δεν θα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις ο πολλαπλασιασμός κοκκίνων γραμμών. γιατί το ίδιο θα κάνουν και οι συνομιλητές μας. Βέβαια επιτρεπτό, θεμητό είναι να επιβεβαιώνουμε και να τονίζουμε τις βασικές μας αρχές όπως αυτή που λέγαμε από την αρχή ε, αυτές ότι τίποτε σε αυτή τη συμφωνία δεν μπορεί να χαμηλώσει το επίπεδο προστασίας του Ευρωπαίου πολίτη εξάλλου και ο πρόεδρος Ομπάμα το ίδιο θέλει για τους Αμερικανούς πολίτες είναι μια κοινή αρχή λοιπόν αυτή επίσης αποσαφηνήσαμε από την αρχή ότι δεν θα διαπραγματευθούμε τίποτε για τις δημόσιες υπηρεσίες και το δικαίωμά μας να αποφασίζουμε αν πρέπει να χορηγείται δημόσια ή ιδιωτικά κάποια υπηρεσία και αυτή είναι μια αρχή που επίσης μάλλον είναι κοινή για τις δύο πλευρές. Όσο θα πλησιάζουμε στην συγγραφή των λεπτομεριών θα αποσαφινιστούν όλα αυτά. Επίσης θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το θέμα των αρνητικών και θετικών καταλόγων. Έχουμε τρία πιθανά πρότυπα. Στη ΣΥΤΑ είναι αρνητικός κατάλογος στον ΚΑΡΤ θετικός και υπάρχει και η πιθανότητα τελικά το TTIP να είναι και θετικό, έχει και θετικό και αρνητικό κατάλογο. το σημαντικότερο είναι ότι όποια και να είναι η προσέγγιση, η αρχή που σας είπα για τις δημόσιες υπηρεσίες θα ισχύσει. Και για μας αυτό είναι το βασικό θέμα. Τέλος, πολλοί από εσά αναρωτήθηκαν αν έχει κανένα επιθετικό συμφέρον η Ένωση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις Παραδείγματος χάριν για τις μη δασμολογικούς φραγμούς και πρόσβαση στην Αμερικανική αγορά. Για το SPS αυτά που ακούστηκαν από τη δική μας πλευρά ίσως ήταν υπερβολικά χλιαρά και αμυντικά, αλλά υπάρχουν και θέματα στα οποία διχτήκαμε πιο επιθετικοί. Όπως σας είπα για τις δημόσιες υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, κινητικότητα και τέλος φυσικά οι προμήθειες είναι βασικό θέμα και από το Κοινοβούλιο θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα σαφή μηνύματα και θέσεις. Θα περιοριστώ σε αυτά γιατί η διαμεσολάβηση των επενδύσεων θα συζητηθεί από την Επίτροπο το απόγευμα και γι' αυτό δεν θα την αναφέρω εγώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Γνάσιο. Επιτρέψτε μου λοιπόν στο τέλος της συζήτησης να αναφέρω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις και να ξεκινήσω με, κάποιες, ε, με κάποια θέματα λεπτομερή και μετά να κοιτάξουμε πιο πολλά θέματα ε, στρατηγικά. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με το θέμα του ISDS. Για να εξηγήσω και πάλι ποια είναι η θέση μου, να πω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και του μέσου που θα χρησιμοποιήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή το γεγονός ότι χρειαζόμαστε μία συμφωνία για τους επενδυτές με τις ίδιες αρχές και την εξίσωση των ε, εγχώριων με τους αλλαταπούς επενδυτές δεν είναι βελτίωση ούτε μειονέκτημα. Αυτό είναι αμφίβολο. Ο κύριος Σιλβάς το, το, το διευκρίνησε ότι τα θέματα των, της επενδυτικής προστασίας είναι θέματα τα οποία σίγουρα θα πρέπει να αναλάβουμε. Το θέμα λοιπόν είναι ποιο εργαλείο είναι το κατάλληλο για να το επιβάλλουμε αυτό. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα και μόνο εργαλείο το οποίο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά περίπτωση τι χρειάζεται. Γιατί στα διάφορα ε, επενδυτικά, σε διάφορες επενδυτικές συμφωνίες έχουμε πολλές διαφορετικές λύσεις και κοιτώντα τι Ηνωμένε Πολιτείε διαπιστώνουμε ότι τα θέματα των διακριτικών μεταχειρήσεων και έχουμε και όλους τους ορισμούς που συνδέονται με αυτό δεν ε, ανακύπτει η Γερμανία έχει 131 συμφωνίες ε, προστασίας επενδύσεων στον κόσμο. Και υπάρχουν μόνο ενδοκρατικές ε, δυνατότητες προστασίας των επενδυτών. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο με μεταξύ της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Αν ε, υπήρχε ανάγκη θα το έχει ζητήσει η γερμανική βιομηχανία. Δεν έχει συμβεί αυτό όμως ως τώρα. Από την άλλη, πρέπει να κοιτάξουμε και τα ποσοστά επενδύσεων των ΗΠΑ σε χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα που έχει τις μεγαλύτερες επενδύσεις από τις ΗΠΑ είναι η Ιρλανδία. Ούτε αυτή η χώρα έχει σύστημα ISDS. Άρα καταφέρνουν αυτές οι χώρες και η Γερμανία και η Ιρλανδία να προστατεύσουν τους επενδυτές χωρίς το σύστημα του ISDS. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι μπορεί να μην χρειάζονται αυτή η στάση. Αλλά η κυρία Ρέντινγκ έχει απόλυτο δίκαιο. Μπορεί να υπάρχουν καταστάσεις όπου να χρειαστεί διαφορετική μορφή προστασία των επενδυτών. Και άρα η συζήτηση αποτελεί ενδεχομένως η συζήτηση για μια διεύρυνση ενός διεθνού οικονομικού δικαστηρίου είναι μια καλή συζήτηση. Το SDS ε, δεν ήταν έως τώρα αγαπητοί συνάδελφοι δικαστήριο με ανεξάρτητους δίκαστες που δεν εξέταζαν ε, τις περιπτώσεις κατά περίπτωση και δεν είχε σαφή κώδικα. Άρα υπάρχουν όλες αυτές οι, όλα αυτά τα θέματα, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε και γι' αυτό λοιπόν η συζήτηση την οποία ξεκινάει ο κύριος Γκάμπριελ, όπως και αυτά που είπε η κυρία Ρέντινγκ, θεωρώ ότι κινούνται προς σωστή κατεύθυνση για το πώς μπορούμε αυτό το παροχημένο ISDS να το εξυγχρονίσουμε, να το πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων της ιστορίας και να δούμε πώς ανεξάρτητα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα δικαστικό όργανο. Κύριε Φιέλνερ, δεν έχετε δίκιο, πιστεύω, δεν είστε σωστά ενημερωμένο σε ό,τι αφορά το θέμα της αντιμετώπισης των επενδύσεων στα πλαίσια της επενδυτικής προστασίας και στο ΣΥΤΑ. Υπάρχει σαφής ρύθμιση ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά από την επένδυση, post-investment. Και ο τομέας ε, εφαρμογής και στο ΣΥΤΑ είναι πολύ περιορισμένο, γιατί θέλουμε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο καταχρήσεων. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αρχή για τις διαπραγματεύσεις με τις ΕΙΠΑ. Κοιτάξτε λοιπόν κύριε Φιέλνερ τι γίνεται με το ΣΥΤΑ. Δεύτερος τομέας, οι υπηρεσίες. Νομίζω ότι αυτό που μόλις είπε ο Ιγνάσιος εκεί και εδώ θα πρέπει να κάτσουμε να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε με σωστό τρόπο τα συμφέροντά μας και κατά πόσον πρέπει να πούμε δογματικά ότι θα πρέπει να ισχύει το ένα ή το άλλο σύστημα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει σημασία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει πρόθεση για τις κοινοφελείς υπηρεσίες που μπορούν να οργανωθούν χωρίς κρατικές επιδοτήσεις. Να προστατεύεται λοιπόν αυτή η αρχή. Να μην τεθεί αυτό ένα αμφιβόλο, αυτό το διτό στοιχείο των υπηρεσιών. Και κατά δεύτερον, γιατί ξαναέθεσε το θέμα της θετικής λίστας. Γιατί υπάρχει όντως το θέμα των νέων υπηρεσιών. Έως τώρα, και είναι σωστό αυτό, ότι η ευρωπαϊκή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η εξή ότι μπορούμε να περιγράψουμε και να ορίσουμε μόνο όσα γνωρίζουμε. Αναγκαστικά. Οι νέε υπηρεσίε θα πρέπει να τύχουν νέα διαπραγμάτευση. Και νομίζω ότι αυτή η αρχή θα πρέπει να προστατευθεί, Γιατί θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε άγνοια σε σχέση με το ποιε υπηρεσίε θα αναπτυχθούν και μετά το άνοιγμα της αγοράς και μετά τις νέες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν. Αυτό λοιπόν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να το εγγυηθούμε, ότι οι νέες υπηρεσίες θα πρέπει να συζητιόνται εκ νέου. Ως εκ τούτου λοιπόν προέκυψε και η σχετική μου πρόταση. για τις τηλεπικοινωνίες και τις τεχνολογίες ε, επικοινωνίας. Θα χαρεί κυρία Ρέντινγκ γιατί έχω να κάνω άλλη μια διευκρίνηση. Ήμουν στο Ανόβερο χτες στην ε, έκθεση ICT και μιλήσαμε επισταμένως με τους εκπρόσωπους ε, της αγοράς για θέματα προσβασιμότητα στην αγορά. Συζητήσαμε το θέμα της μη ρύθμισης στις επαφές με και το κατά πόσον υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Θα πρέπει να εκφράσουμε το δημόσιο συμφέρον το δικό μας. σε ό,τι αφορά και την ανάπτυξη κοινών προτύπων για να αποφύγουμε διακριτική μεταχείριση. Όλα αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν λοιπόν και φυσικά σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτών στα, στα πλαίσια του e-commerce, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα πρέπει να κάνουμε σαφείς διατυπώσεις. Και τα λοιπόν ανακύπτει και το ερώτημα της προστασίας των δεδομένων. Και εδώ συμφωνώ με τους συναδέλφους που λένε ότι χρειαζόμαστε τάχιστα την ψήφιση του βασικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων για να ξέρουμε με σαφήνεια πώς θα διασφαλιστεί το δικό μας επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Ήταν καθοριστικό θέμα αυτό και στη συζήτηση με τους συναδέλφους στην έκθεση χτες ότι θα πρέπει να πρόκειται για ένα κανονισμό ο οποίος θα ισχύει εξίσου σε όλες τις ε, ε, ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση διαφορετικά πρότυπα στις διάφορες χώρες και πόσο μάλλον και στη Γερμανία διαφορετική ισχύ ανάλογα με το κρατήδιο. Αυτό αγαπητοί συνάδελφοι είναι προς το συμφέρον και των Αμερικανών παρόχων λογισμικού να υπάρχει ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο για την προστασία των δεδομένων. Τρίτος τομέας, το θέμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εδώ όντως πιστεύω ότι αν ένα, μια τέτοια εμπορική συμφωνία ε, θα πρέπει να ανοίξει τον ανταγωνισμό, θα πρέπει να είναι και δίκαιος ο ανταγωνισμός αυτός. Γιατί ε, με τη μείωση των εμπορικών φραγμών θα έχουμε πιο μεγάλη ανταγωνιστικότητα και θα πρέπει αυτό να βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Να βασίζεται στην αποδοτικότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων και όχι σε θέματα κοινωνικού ντάμπινγκ. Γι' αυτό λοιπόν για μένα προσωπικά το θέμα ενός βασικού όγκου ο εργασιακού δικαίου είναι κρίσιμο για να μην υπάρξει κοινωνικό dumping. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε αυτά. Επισταμένος. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Στην εσωτερική αγορά μεταξύ Φιλανδίας και Σικελίας και Πορτογαλίας και Λιτωνίας υπάρχουν ε, διαφορετικά πρότυπα, δεν υπάρχουν. Ε. Τι θέλουμε λοιπόν. Πώς θα αποδεχτούμε λοιπόν, πώς αποδεχόμαστε την ενιαία αγορά και είμαστε ικανοποιημένοι με την ενιαία αγορά. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι σαφές λέει ο Πρόεδρος ότι δεν θέλουμε να μεταφέρουμε το εργασιακό δικαίωμα του Λουξεμβούργου στις ΗΠΑ. Μιλάμε για βασικές αρχές οι οποίες ισχύουν και σε άλλες εμπορικές ε, συμφωνίες που έχουμε συνάψει. τα οποία τα θέτουν και άλλοι εμπορικοί εταίροι του πλανήτη. Δεν απαντάει ο πρόεδρος. Είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό, δεν λέω. Επειδή έχουμε και παραδείγματα όπου προέκυψαν με τον τρόπο αυτό ανταγωνιστικά πλέον εκτήματα. Το θέμα επίσης που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι κοιτώντας τις ευρωπαϊκές εταιρείες... που στην Ευρώπη κάνουν συναλλαγές κοινωνικές και έχουν εγκατασταθεί στα νότιε πολιτείε των ΗΠΑ και εκεί ε, λειτουργούν χωρίς καν συνδικάτα. Είναι ελκυστικό ο τρόπο λειτουργίας αυτό αναρωτιέμαι. Ναι. Η σωστή η κανονιστική, η ρυθμιστική συνεργασία. Το θέμα αυτό τέθηκε. Νομίζω ότι τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί, όπως η ομάδα εργασίας υπαριθμών 29, νομίζω ότι μπορούν να εξετάσουν τα πρότυπα τα οποία θα κληθούν να εγκρίνουν τα κοινοβούλια. Μπορούμε να αναπτύξουμε λοιπόν το μοντέλο αυτό και να δούμε τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε για να διευκρινίσουμε τα κείμενα τα διαπραγματευτικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αυτό τέθηκε ως θέμα Νομίζω ότι πρόκειται για μεγάλο συμφέρον από δική μας πλευρά. Θα πρέπει να υπάρχει σαφή διατύπωση στα πλαίσια του G20 για να υπάρχει σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτά είναι κάποια μεμονωμένα στοιχεία μόνο, τα οποία όμως κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, την οποία ανέφεραν και κάποιοι συνάδελφοι. Να διατυπώσουμε με επιθετικό τρόπο τις ευρωπαϊκές μας θέσεις. Και αυτό προσπάθησα να κάνω στην έκθεσή μου. Γιατί πιστεύω Έχουμε κάποιες αντιλήψεις για την κοινωνία και θα πρέπει να τις εξαγάγουμε αυτές τις ε, ιδέε και να δώσουμε λίγη έμφαση εν των Ηνωμένων Εθνών, των Ηνωμένων Πολιτειών, Γιατί το επίπεδο της ε, προθυμίας δεν βλέπω να έχει κινηθεί ιδιαίτερω. για την διαδικασία fast track, για το TPA. Φαίνεται ότι προκαλεί μεγάλη διαφωνία. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πού θέλουμε να κατευθυνθούμε εμείς. Πώς θέλουμε εμείς να διαμορφωθεί μια εμπορική συμφωνία. Ως εκ τούτου. Νομίζω ότι μετά από 1,5 χρόνο διαπραγματεύσεων και συζητήσεων είναι λογικό να εξετάσει το Κοινοβούλιο την κατάσταση και να κάνει έναν απολογισμό. και ίσως με φρέσκο μάτι να ξεκινήσουμε τη δουλειά εκ νέου για να προαγάγουμε τα ευρωπαϊκά μας εμφέροντα. Και φυσικά είναι σημαντικό προς την κατεύθυνση αυτή να αναπτύξουμε μια κοινή τοποθέτηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί θέλω να αποφύγω στο τελική ανάλυση να είναι οριακά τα αποτελέσματα στην ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Ας προσπαθήσουμε να το αποφατηθούμε με κοινό τρόπο για να έχουμε μία επιθετική προέθηση των ε, συμφερόντων μας, των προτύπων μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι με μεγάλη προσοχή θα εξετάσω τις τροπολογίες σας, θα κάνω προτάσεις συμβιβαστικές και τις γνωμοδοτήσεις των ε, άλλων επιτροπών. Σας υπενθυμίζω ότι είναι 14 οι επιτροπές που γνωμοδοτούν. Αυτό δεν έχει επαναληφθεί ποτέ στην ιστορία του Κοινοβουλίου. Και αυτό γιατί προφανώς θα πρέπει να κοιτάξουμε τον τομέα αρμοδοτήτη των ε, των διαφορών επιτροπών που θα επισημάνουν στοιχεία τα οποία δεν έχουμε λάβει υπόψη. 26 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία ναι. κατάθεση τροπολογιών. Για να παρουσιάσετε τις αντιλήψεις σας και να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας με όσο πιο συνεκτικό τρόπο γίνεται για να καταρτήσουμε και μια συνεκτική έκθεση τελική ανάλυση. Στην Επιτροπή θα ψηφίσουμε 6 Μαΐου και στην Ολομέλεια μεταξύ 18 και 21 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολυάριθμες παρεμβάσεις και προσβλέπω στη μελλοντική επικοδομητική συζήτηση. Στις 11.30 έχουμε συνάντηση των συντονιστών.